Πρόεδρο. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθεί να αρχίσει η συνεδρίαση αυτή στην ώρα της. Λοιπόν, καλωσορίζω όλους στην συνάντηση αυτή με τον οριστέντα Επίτροπο, κύριο Γιάννης Λενάρτσης, ο οποίος είναι υπεύθυνο για την ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική προστασία διαχείριση κρίσεων. Ερωτήσεις θα υποβάλουν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και από την Επιτροπή ΔΕΒΕ. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι συνδεδεμένη επιτροπή. Και πριν να αρχίσουμε θα ήθελα να σας παρακαλώ να σας πω τα τυπικά. Τι ισχύει δηλαδή για αυτήν την ακρόαση. Σας υπενθυμίζω πρώτα απ' όλα ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί τους οριστέντες επιτρόπους βάσει των γενικών τους ικανοτήτων της ε, δέσμευσής τους υπέρ της Ευρώπης και της προσωπικής τους ανεξαρτησίας. Επίσης, αξιολογεί τις γνώσεις τους, τις σχετικές με το χαρτοφυλάκιο το οποίο αναλαμβάνουν και τις ικανότητες επικοινωνίας που έχουν. Υπερθυμίζω επίσης ότι πριν από την ακρόαση, ο οριστής επίτροπος έχει απαντήσει γραπτά σε διάφορες ερωτήσεις που έχουμε υποβάλει επίσης γραπτά. Και αυτέ οι απαντήσει έχουν μοιραστεί σε όλες τι γλώσσες. Υπενθυμίζω ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δεν έχει γύρει καμία ένσταση για την διεξαγωγή της ακρόασης αυτής. Επιθυμίζω επίσης, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ε, η Δημόσια υγεία και Ασφάλειας είναι συνδεδεμένη επιτροπή σε αυτή την ακρόαση. Τώρα θα σας εξηγήσω τα πρακτικά. Ότι ο οριστής επίτροπος καλείται να κάνει μια αρχική παρουσίαση 15 λεπτών. Επίσης, το τέλος της ακρόασης έχει στη διάθεσή του άλλα 5 λεπτά. Εισαγωγικά θα ακούσουμε 25 ερωτήσεις από ευρωβουλευτές. Η συζήτηση θα λάβει η χώρα ως εξής. 5 λεπτά αρχικά ε, έχει στη διάθεσή του ο καθένα για ερώτηση και απάντηση, ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση και εφόσον υπάρξει και δεύτερη ερώτηση από τον ίδιο βουλευτή, έχει στη διάθεσή του ένα λεπτό και ένα λεπτό θα κρατήσει και η απάντηση. Ο πρώτος γύρος θα αποτελείται από 7 ερωτήσεις που θα θέσουν διάφορες πολιτικές ομάδες. Στο δεύτερο γύρο θα έχουμε 18 ερωτήσεις ε, που βασίζονται γενικά στην κατανομή μεταξύ των πολιτικών ομάδων και θα συμπεριληφθούν εκεί και ε, μέλη μη εγγεγραμμένοι. Θέλω επίσης, συνάδελφοι, να σας υπενθυμίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρείτε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε διερμηνία σήμερα σε 23 γλώσσες. Μπορείτε λοιπόν να μιλήσετε στην δική σας τη μητρική γλώσσα. Μην ξεχνάτε όμως ότι πρέπει να μιλάτε, σίγα να μην μιλάτε πολύ γρήγορα έτσι ώστε να μεταφραστούν όλα τέλεια. Επίσης, μην ξεχνάτε όταν μιλάτε και υποβάλλετε την ερώτησή σας να μην κρατάτε τα ακουστικά στα αυτιά σας, να τα απομακρύνετε από το μικρόφωνο παρακαλώ. Επίσης σας πληροφορώ ότι η συζήτηση αυτή αναμεταδίδεται live ε, στο διαδίκτυο και επίσης μπορείτε και αργότερα αν θέλετε ε, να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένα την συνάντηση αυτή. Και πάλι λοιπόν ε, σας καλωσορίζουμε εδώ στην Επιτροπή μας, κύριο Ριστέντα Επίτροπο. Πριν σας δώσω το λόγο, απλώς θέλω να τονίσω πόσο μεγάλη σημασία έχει το χαρτοφυλάκιό σας για την Επιτροπή μας. Και θέλω επίσης να πω ότι ελπίζω να έχουμε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας, εφόσον αναλάβετε τα καθήκοντά σας. Το χαρτοφυλάκιό σα, δηλαδή ανθρωπιστική βοήθεια, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την Επιτροπή ανάπτυξη, γιατί οι ανθρωπιστικές κρίσεις γίνονται όλο και συχνότερες, κρατάνε περισσότερο και είναι και πιο περίπλοκες. Έχουμε και την κλιματική αλλαγή μεταξύ άλλων. Οι ανθρωπιστικοί πόροι ποτέ δεν θα φτάνουν βέβαια, αλλά εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει αρκετή ανθρωπιστική χρηματοδότηση και ότι ε, προσφέρονται τα κονδύλια με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί διεθνώς όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια τα τελευταία χρόνια και τώρα όλα αυτά τίθενται σε εφαρμογή από τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε προσβλέπουμε να ακούσουμε τον οριστέντε επίτροπο σήμερα, να μάθουμε πώς θα προχωρήσετε στο έργο σας βάσει των δεσμεύσεων που έχουν αναλυθεί στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής προστασίας και πώς όλα αυτά ε, θα τα βάλετε στο αυλάκι και τι ρόλο επιφυλάσσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλα αυτά. Οπότε, κύριε Λινάτσης, για άλλη μια φορά σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας και έχετε το λόγο παρακαλώ για 15 λεπτά. Αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, είναι διπλή τιμή για αυτή για μένα. Καταρχάς που είμαι υποψήφιος της Σλοβενίας για είναι με στο μέλος του επομένου σώματος της ε, Κομισιόν. Και μετά, εάν συμφωνήσετε εσείς, θα αναλάβω την ευθύνη της ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής προστασίας στα πλαίσια της διαχείρισης των κρίσεων. Σαν Σλοβαίνος μπορώ να κατανοήσω απόλυτα το γεγονός ότι σήμερα αυτό που είναι η Γενική Διεύθυνση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία και τις διάφορες επιχείρησεις ανθρωπιστική βοήθεια δημιουργήθηκε το 1992 Επίσης ήταν μια ανταπόκριση στους πολέμους στην επικράτεια της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Τον ίδιο χρόνο η αρμοστία του ΟΗΕ για τους ε, πρόσφυγες δημιουργήσε ένα, μια υπηρεσία, ένα γραφείο στη Σλοβενία. Πριν να αποφυτίσω από τη νομική και εγώ συμμετείχα ήθελα να τους βοηθήσω να φροντίσουν για τους πρόσφυγες που έφευγαν ή περνούσαν από τη Σλοβενία. Αυτό με έδωσε δυνατότητα για την πρώτη μου ε, μετριοπαθή συνεισφορά στην ανθρωπιστικό έργο. Μετά από 25 χρόνια είμαι μπροστά σας σαν υποψήφιος επίτροπος. Εάν μου ανατεθεί αυτό το καθήκον, σας διαβεβαιώνω ότι θα αφιερώσω όλη μου την ενέργεια και σχεδόν τρεις δεκαετίες εμπειρίας σε διεθνή και ευρωπαϊκά βήματα συζητήσεων να βοηθήσω να, μειωθεί, να μειωθούν τα δεινά και να δώσω ανακούφιση στους ανθρώπους που πλήττονται από κρίσεις και έτσι θα παγιώσω και θα βεβαιώσω την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, μια αξία στην οποία ένθερμα πιστεύω. Αξιότιμα μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζεται ευρέω σαν υπεύθυνο ηγέτη σε παγκόσμιο προσκήνιο για ανθρωπιστική βοήθεια και θέλουμε, πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Όμω, για να ενισχύσουμε αυτό το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναβαθμίσει τι δυνατότητε που έχει για να μπορεί να βοηθήσει περισσότερου ανθρώπου που έχουν ανάγκη με αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο. Επί του παρόντο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, καλύπτει περίπου 100 εκατομμύρια ανθρώπου που έχουν ανάγκη κάθε χρόνο. Του βοηθούμε αυτού και εντό και εκτό τη Ένωση. Αυτό επηρεάζει άμεσα τι ζωέ ανδρών, γυναικών και παιδιών χωρί διάκριση βάσει τη εθνικότητά του. Τη φιλής του, του φίλου του, θρησκευτικών πεπιθέσεων, τάξεω ή πολιτικών απόψεων. Είναι καθησυχαστικό να σημειώνει κανείς ότι περίπου 90% από τους Ευρωπαίους υποστηρίζουν τη δράση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής προστασίας. Επίσης γνωρίζω ότι αυτές οι προσπάθειες παραδοσιακά απολάμβαναν ισχυρή υποστήριξη από το Κοινοβούλιο. Σας διαβεβαιώνω ότι έχω κάθε πρόθεση να συνεργαστώ μαζί σας, να σας ενημερώνω, να σας τηρώ ενήμερους και να ακούσω τις απόψεις σας και τις ανησυχίες σας. Αξιότιμα μέλη, αυτός ο διορισμός μου σημαίνει μια εξαιρετική δυνατότητα και ευκαιρία να υπηρετήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχω επίγνωση των πολλαπλών προβλημάτων και ε, προκλήσεων που αντιμετωπίζει αυτό το χαρτοφυλάκιο διαχειρίσεω κρίσεων. Σήμερα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Σχεδόν 71 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίζονται βία και όχι μόνο λόγω συγκρούσεων. Κάθε χρόνο, περίπου 70.000 άνθρωποι πεθαίνουν και άλλα 70 εκατομμύρια άνθρωποι τραυματίζονται και μένουν άστεγοι ή χρειάζονται κατεπίγουσα βοήθεια σαν αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών. Δίπλα σε αυτά τα θύματα ε, έχουμε και το κόστος που είναι πολύ ψηλό και εξακολουθεί να αυξάνεται. Από το 2010 οι φυσικές καταστροφές έχουν προκαλέσει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ σε ζημίες κάθε χρόνο και μόνο στην Ευρώπη αυτό. Ε, ακόμα χειρότερα, οι τάσεις που αντιμετωπίζουμε είναι ανησυχητικέ. Οι ανθρωπιστικές κρίσεις διαρκούν περισσότερο και είναι περιπλοκότερες από ό,τι κατά το παρελθόν. Οι φυσικέ και ανθρωπογενεί καταστροφέ συμβαίνουν με αυξανόμενη συχνότητα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι πλήττονται και στην Ευρώπη. Μέχρι το 2050 θα, ίσως θα έχουμε πάνω από 140 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους στην υποσαχάρια Αφρική, την Νότια Ασία και τη Λατινική Αμερική. Πόσοι από αυτούς θα μπορέσουν να ξαναβρούν αυτά που τους έχουν απομείνει και να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη ή σε άλλα μέρη για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Οι παγκόσμια διαθέσιμοι πόροι για τη διαχείριση των κρίσεων δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες, ούτε καν βέβαια στις μελλοντικέ προβλεπόμενες. Υπάρχει ένα κενό διευρυνόμενο όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα έχουμε την αλλαγή του κλίματος που αλλάζει το, τοπίο, αλλαγή του κλίματος και αυξάνει τις, υφιστάμενες, αυξάνει τις υφιστάμενες εντάσεις. Σε κάθε έκθεση μαθαίνουν περισσότερο για την αλλαγή του κλίματος και τον αντίκτυπο που έχει αύξηση του, του των θαλασσών, ε, αυξάνεται η ένταση των καταιγίδων, ε, περισσότερες περιόδους, μακρύτερες περιόδους ξηρασίας, καταστροφικές πλημμύρες και τα οικοσυστήματα πάσχουν. Χρειαζόμαστε άλλη μια έκθεση για να πιστούμε ότι είναι σοβαρή αυτή η αλλαγή του κλίματος. Η νέα γενιά σίγουρα και προφανώς ε, δεν χρειάζεται άλλη έκθεση. Ξέρει πολύ καλά ότι το σπίτι μας καίγεται για να χειροτερέψουμε τα πράγματα, ποια μέρη του κόσμου που πλήττονται από τις αλλαγές του κλίματος σκληρότερα είναι και οι πιο έφταστες και οι λιγότερο ανθεκτικές περιοχές, όπως οι χώρες του Σαχέλ και του κέρατος της Αφρικής, για να παραθέσω μόνο δύο παραδείγματα. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσω σαν Επίτροπος για Διαχείριση των Κρίσεων. Καταλαβαίνω ότι η εικόνα που ζωγράφισα είναι ζωφερή, αλλά δεν παρετούμε και μάλιστα βλέπω αυτές τις προκλήσεις που περιέγραψα και σαν ευκαιρίες. Ευκαιρίες να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα και με διαφορετικό τρόπο να βασιστούμε στα, σε αυτά που λειτουργούν καλά και να διορθώσουμε αυτό που δεν λειτουργεί καλά. Επίσης καταλαβαίνω ότι ποικιλοτρόπως μπορώ να είμαι ευγνώμων για την αποφασιστικότητα και επιτεύγματα των προκατόχων μου που είχαν μεγάλα κίνητρα, το προσωπικό της DG ECO, τους διεθνείς εταίρους και πιο σημαντικά τους διάφορους εργαζόμενους στον τομέα της ανακούφισης των πληγέντων. Λόγω των ακαμάτων προσπαθειών τους ε, ε, τα πράγματα ε, βελτιώνονται. Επίσης είναι σεβαστή, γίνεται σεβαστή η Ευρωπαϊκή Ένωση διότι είναι προσκολλημένη στις βασικές ανθρωπιστικές της αρχές. Ανθρωπισμού, ουδετερότητα, μεροληψία και ανεξαρτησία. Εγώ θα υπερασπιστώ αυτές τις αρχές στο μέλλον. Τώρα στρέφομαι προς τις προτεραιότητες που έχω καθορίσει, αν τελικά επιβεβαιωθεί ο διορισμό μου σαν Επίτροπο Διαχείριση των Κρίσεων και σαν, σαν Ευρωπαίο Συντονιστή για την ανταπόκριση στι κατεπήγουσε ανάγκε, θα υποστηρίξω αυτού που έχουν ανάγκη όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά γίνεται, σεβόμενο πλήρω τι αρχέ τι ανθρωπιστικέ. Σχετικά με αυτό, θα μεγιστοποιήσω την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα τη ανταπόκρισή μα στι κρίσει, ούτω ώστε να καλύπτουμε όσο δυνατόν περισσότερου ανθρώπου που έχουν ανάγκη. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε καλύτερα σύμφωνα με την δοθήσα εντολή. Προτίθεμαι να ενισχύσω το, το, κέντρο συντονισμού για ανταπόκριση τη κρίση Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορεί να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπίσει διάφορε κρίσει, ευρύ φάσμα. Ακόμα πολύ σημαντικό, αν επιβεβαιωθώ, θα εστιαστώ στο να προωθώ σε παγκόσμιο προσκήνιο την, το, διεθνή, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Λοιπόν, θα, σε όλους τους φορείς θα τονίσω την ανάγκη να υπάρχει ανθρωπιστικός χώρος. Είναι απαράδεκτο ότι οι ανθρωπιστικοί φορείς όλο και περισσότερο είναι στόχοι και η πρόσβασή τους στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη ε, μπλοκάρεται πάρα πολύ συχνά και τακτικά. Δεύτερον, σύμφωνα με την προτινόμενη εντολή, θα εντατικοποιήσω τι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να προλάβει τι καταστροφέ και να μην συμβαίνουν εν πρώτη. Επίση, να ενισχύσω και τη δυνατότητα που θα έχουμε να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Λαμβάνοντα υπόψη προβολέ για την αλλαγή του κλίματο, παρατεταμένε συγκρούσει και αυξανόμενη αστάθεια σε όλο τον κόσμο, εμεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αυτή, πρέπει να εργαστούμε με έναν ολοκληρωμένο τρόπο Εάν δεν το κάνουμε αυτό, θα υπονομεύσουμε την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, που είναι συλλογική ευθύνη. Σχετικά με αυτό, καλωσορίζω την προσέγγιση που εξετάζει η ενεκλεγήσα πρόεδρος. Σύμφωνα με αυτήν, ο κάθε επίτροπος πρέπει να εξασφαλίζει ότι θα πρέπει να επιτευχθούν οι διάφοροι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης στους αντίστοιχους τομείς. Πέρα από την πρόληψη, προτίθεμαι να συνεργαστώ στενά με την είπατε εκπρόσωπο, αντιπρόεδρο και άλλα μέλη του κολεγίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα είναι υπεύθυνοι για τομείς όπως είναι η αλλαγή του κλίματος, το περιβάλλον και η ανάπτυξη. Στόχος είναι να εξασφαλίσουμε ότι η μείωση του κινδύνου καταστροφών θα είναι ένα απόσπαστο τμήμα των προσπαθειών που θα καταβάλουμε να αυξήσουμε την αντοχή των κοινωνιών μας και των οικοσυστημάτων μας, ξεκινώντας από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αξιότιμα μέλη, η ανθρωπιστική βοήθεια και ανταπόκριση καταστροφέ πρέπει να ειδωθεί ότι είναι ένα εργαλείο τη τελευταία ε, γραμμή, αν θέλετε, το έσχατο μέσο, όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει. Το να αποφύγουμε μια τέτοια αποτυχία πρέπει να είναι η πρώτη μας ε, μέρημνα. Όταν πρέπει να κινητοποιήσουμε ανθρωπιστική βοήθεια, στόχος θα πρέπει να είναι να εξαρτηθούμε από αυτή τη βοήθεια για το βραχύτερο δυνατόν διάστημα. Με άλλα λόγια, πρέπει οι άνθρωποι να βγουν από το χώρο των, των για να μπορέσουν να κτίσουν τις δυνάμεις τους και να μπορέσουν να ωφεληθούν από μακροπρόθεσμες βιώσιμες λύσεις. Εδώ η ασφάλεια και η ανάπτυξη και οι σχετικές πολιτικές, ε, παίζουν ιδιαίτερο ρόλο. Σε έφταστες χώρες, κυρίως εκείνες οι οποίες περνάνε από παρατεταμένες κρίσεις, θα πρέπει να εργαστούμε προς ανθρωπιστικό κόμβο ε, που θα συγκεράσει ανάπτυξη και ειρήνη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι τοπικέ ιδιαιτερότητε και να δώσουμε την καλύτερη βοήθεια σε αυτού που έχουν την ανάγκη, προσέχοντα ιδιαίτερα βέβαια τις πλέον ευάλωτε ομάδες όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Αυτό θα απαιτήσει νέε συνεργασίες, επίσης και καινοτόμα εργαλεία εδώ ιδιαίτερα θα ήθελα να κάνω περισσότερα ούτω ώστε να ενισχύσω τοπικού φορεί στην επίδοση επιτόπια βοήθεια, Γνωρίζουν καλύτερα το όλο πλαίσιο, μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικότερα και γνωρίζουν τι ε, έχει αποτέλεσμα και τι δεν έχει. Ταυτόχρονα όλοι γνωρίζουμε ότι παρά τι προσπάθειε δεν μπορούμε να αποφύγουμε τα πάντα. Πρόσφατα γεγονότα συμπεριλαμβανομένε των ε, θανατηφόρων πυρκαγιών στην Πορτογαλία των προσφάτων Αυτά έχουν δείξει ότι πρέπει να βελτιωθούμε όσον αφορά την αποφυγή των καταστροφών και θα πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να μπορούμε να ανταποκριθούμε όταν η πρόληψη έχει αποτύχει. Γι' αυτό προτίθαμε να επιδιώξω ένθερμα ενισχυμένη εφαρμογή του Rescue, δηλαδή τον ενισχυμένο μηχανισμό πολιτική προστασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε ενισχυμένε δυνατότητε για να αντιμετωπίσουμε τι δασικέ πυρκαγιέ, κατεπίγουσες ιατρικέ ανάγκες, χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές καταστροφές. Εδώ πρέπει να πω ότι βασίζομαι στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτω ώστε αυτό να μπορέσει πραγματικά να υλοποιηθεί και να γίνει πραγματικότητα. Τρίτη προτεραιότητα, θα πρέπει να αυξήσουμε την ορατότητα του τρόπου που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση τη κρίση. Θα βασιστώ στην ισχυρή υποστήριξη που ήδη απολαμβάνει η ανθρωπιστική βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ενώση από πλευρά Ευρωπαίων πολιτών. Και θέλω να διαβεβαιώσω του πολίτε ότι κάθε ευρώ που δαπανάτε σε αυτό το τομέα είναι ένα ευρώ που ξοδεύεται σωστά. Το πιο σημαντικό ακροατήριο θα πρέπει να είναι οι πολίτε και οι δικαιούχοι τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Γι' αυτό θα θέσω υψίστη προτεραιότητα στο θέμα τη επικοινωνία με αυτού. Αξιότιμα μέλη, δεν θα κρύψω το γεγονός ότι αυτές οι προτεραιότητες και αυτοί οι στόχοι έχουν ένα κόστος. Αλλά αντί να μιλάω για κόστος και δαπάνες, θα προτιμούσα να μιλήσω για επενδύσεις. Εν τη αυτή περιπτώσει, επένδυση στο κοινό μας μέλλον. Γι' αυτό σας καλώ για την υποστήριξή σας. Να εξασφαλίσουμε την προτινόμενη αύξηση του 30% του προϋπολογισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια σαν ένα τμήμα του νέου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό είναι σημαντικό ούτω ώστε να πετύχουμε του στόχου που έχουμε θέσει που είναι φιλόδοξοι την επόμενη πενταετία και πέρα από αυτή την πενταετία. Επίση, εκτιμούσα τη συνεχιζόμενη υποστήριξή σα, εξασφαλίζουμε αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των πόρων. Από την πλευρά μου, σα εγγυώμαι ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να χορηγείται σε αυτού που χρειάζονται διαφανώ και βάσει υγιού ε, δημοσιονομική διαχείριση. Εκτελώντα τα καθήκοντά μου, θα είμαι έτοιμο να συνεργαστώ στενά και με τις δύο επιτροπές που είναι εδώ παρούσες. Εάν πετύχω να κερδίσω την εμπιστοσύνη σας, θα ήθελα να, να δούμε πίσω μετά από πέντε χρόνια και να δούμε ότι κάναμε τη διαφορά. Ότι έχουμε βοηθήσει να ανακουφίσουμε το μαρτύριο, τα προβλήματα πολλών, ότι έχουμε συμβάλει στη δημιουργία πιο ανθεκτικών κοινοτήτων και ανθρώπων για ένα φυσικό περιβάλλον που είναι υγιέστερο και πιο ανθεκτικό και να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο μέλλον τους οι Ευρωπαίοι. Σας ευχαριστώ. Thank you for... Uh, σας ευχαριστώ για τα εισαγωγικά σας σχόλια, κύριε υποψήφιο Επιτροπέ. Και τώρα να ξεκινήσουμε τον πρώτο γύρο με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Να δώσω το λόγο στο Γιώργη Χόλβανη από το ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Και θα συνεχίσω στα, στη μητρική μου γλώσσα, αν θέλετε να βάλετε τα ακουστικά σας. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία μας έδωσε η Πατή του ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2019 186.600 Σύριοι πρόσφυγες ε, επέστρεψαν στη Συρία από την Αίγυπτο, το Ιράκ και άλλες χώρες μεταξύ το... μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Παρά το γεγονό ότι δεν υπάρχει ακόμα ειρήνη στην Συρία, υπάρχουν ε, ενδείξεις ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την αναμόρφωση της χώρας. Και πολλοί από τους πρόσφυγες λοιπόν αποφάσισαν να επιστρέψουν τους επόμενους μήνες. Το πρόβλημα των 6 εκατομμυρίων περίπου ε, εσωτερικά εκτοπιστέντων θα πρέπει επίσης να επληθεί. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να συνεχίσουν τις ζωές τους στην ε, χώρα των ε, προγόνων τους. Είναι τρομερές οι διώξεις από το Ισλαμικό κράτος. Θα πρέπει να τους δώσουμε ό,τι βοήθεια μπορούμε. Μετά από 8 και πλέον έτη πολέμου, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται κάποιες βασικές υπηρεσίες, κάποιες βασικές υποδομές, πόσιμο νερό, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση. Προκειμένου λοιπόν οι Σύριοι να μπορέσουν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα παραμονή στην πατρίδα του, θα πρέπει να υπάρχουν αυτέ οι βασικέ προποθέσει. Δεδομένου λοιπόν του πλαισίου αυτού, κύριε υποψήφια Επιτροπέ, πώς σκοπεύετε να βοηθήσετε τους ήρους μετανάστες και να καλύψετε τις ανθρωπιστικές τους ανάγκες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει ο Πρόεδρος να επενθυμίσω ότι θα πρέπει να τηρήσουμε το ένα λεπτό χρόνο που προβλέπετε. Ξεπεράσατε το λεπτό σας. Να δώσω το λόγο όμως στον υποψήφιο Επιτροπό για να απαντήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε για την ερώτηση αυτή. Θα, ακούσω, θα ακολουθήσω την δηλωμένη μας αρχή σε ό,τι αφορά τις επιστροφές. Αυτό σημαίνει ότι θα υποστηρίξουμε και θα προωθήσουμε τις επιστροφές που είναι ασφαλείς, με αξιοπρέπεια και είναι και βιώσιμες. Και ακόμα πιο σημαντικό, εθελούσιες. Προς το παρόν, η εκτίμησή μου είναι ότι οι συνθήκες αυτές ακόμα δεν συντρέχουν στη Συρία. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου να γίνουν αυτές οι επιστροφές. Και συμφωνώ μαζί σας απόλυτα ότι η ανοικοδόμηση της Συρίας θα σημαίνει τεράστιες, μα τεράστιες επενδύσεις. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό. Για προφανείς λόγους. Επίσης, ε, δεν πληρούνται και προποθέσει ό,τι αφορά και άλλα μέσα και εργαλεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξεχνάμε τους εσωτερικά εκτοπιστέντε στην Συρία, στο εσωτερικό της Συρία. Η Επιτροπή, μάλιστα, παρέχει το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας στους ανθρώπους αυτούς μέσω των γειτονικών χωρών και μέσω τη Δαμασκού. Παρέχοντα λοιπόν την ανθρωπιστική αυτή βοήθεια για του ιστορικά εκτοπιστέντε και για τους πρόσφυγες τη Συρίας, δεν κάνουμε διάκριση βάσει των θρησκευτικών πεπιθήσεων, βάσει και των αρχών τι οποίε ανέφερα στα εισαγωγικά μου σχόλια σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια προ ε, τέτοιου λαού, Υπάρχει αυτή η αρχή τη αμεροληψία, την οποία και σκοπεύω να προασπιστώ με στένος. Αυτή η αρχή συνεπάγεται ότι η ανθρωπιστική βοήθεια χορηγείται εκεί που χρειάζεται πιο πολύ, χωρί να λαμβάνουμε υπόψη προσωπικά χαρακτηριστικά, στα οποία συγκαταλέγεται και η θρησκεία. Να σας ε, διαβεβαιώσω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει και βοηθά και μέλη χριστιανικών ε, κοινοτήτων που έχουν υποστεί διώξεις, που έχουν ε, είναι πρόσφυγες και αυτό και στην Συρία αλλά και στο Ιράκ, στο Βόρειο Ιράκ. Ευχαριστώ πολύ. Συμπληρωματική ερώτηση τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας αυτή. Αντιμετωπίσουμε ακόμα μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις στην Αφρική, όπου οι θρησκευτικέ και εθνοτικέ συγκρούσει ε, θα μπορούσαν να προκαλέσουν ε, νέε ανθρωπιστικέ ε, αιστείε προβλημάτων. Συμφωνείτε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρώπη πρέπει να ακολουθεί την αρχή του ότι χορηγείται εκεί που χρειάζεται πιο πολύ ή θα ακολουθήσετε τις καλές πρακτικές των ιδρυμάτων των κρατών μελών. Δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα αξιότιμη κυρία Βουλευτά την ερώτησή σας ε, σωστά και ζητώ συγγνώμη. Αλλά και στην Αφρική εξίσου θα επιμείνω η ανθρωπιστική βοήθεια να χορηγηθεί σε αυτούς που τη χρειάζονται πιο πολύ βάσει των αρχών της αμεροληψίας. Δίνουμε βοήθεια σε όποιον τη χρειάζεται. Προς τη διαδικασία αυτή στηριζόμαστε στους εταίρους μας από τον ΟΗΕ, η UNICEF για παράδειγμα, η πατερμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, το πρόγραμμα του World Food και επίσης σε ένα μεγάλο βαθμό και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις μας ε, που έχουμε δώσει, θα επιμείνω και στη χορήγηση βοήθειας και στου τοπικού φορείς. Όπως είπα και εισαγωγικά, αυτοί είναι που γνωρίζουν σε βάθος τι γίνεται επί τόπου, αυτοί είναι εκείνοι που μπορούν να δώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριο Νόμπερτ Νόιζερ. Παρακαλώ. Καλώς ήρθατε. Και σας ευχαριστώ πολύ κύριε οριστέντα επίτροπη. Η ερώτηση σας έρχεται από πίσω, από την πλάτη. Δεν είναι επικίνδυνο όμως η ερώτηση. Και θα συνεχίσω γερμανικά. Στην δήλωσή σας είπατε ότι υπάρχουν ε, διάφορες πηγές ε, φυσικών καταστροφών και ε, συγκρούσεων. Χρειάζεται λοιπόν κατεπίγουσα βοήθεια και χρειαζόμαστε επίσης μια ευέλικτη δικτύωση με το σκέλος της ε, πολιτικής ε, βοήθειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Γιατί πολλές χώρες δεν μπορούν να παρέχουν αυτές τις βασικές υπηρεσίες στους λαούς τους. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει οι πολίτες να εμπλακούν σε όλη αυτή τη διαδικασία και έχουμε τη σχέση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής βοήθειας. Ως νέος επιτροπός λοιπόν πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε αυτή τη σύνδεση και πώς κρίνετε την προσέγγιση σε διπλωτικά προγράμματα όπως ε, στο Τσάντ, Νιγηρία ε, και Ουγκάντα και στο Τσάντ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμη Ευρωβουλευτά. Ναι, είναι ευτυχώ γυρνάει η καρέκλα, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα αν η ερώτηση μου έρχεται από την πλάτη. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Θέλω να υπογραμμίσω ότι οι δραστηριότητές μας ανθρωπιστικής βοήθειας ε, συμπληρώνονται με τις, και είναι απόλυτα συμβατές ε, με τις δράσεις μας για την προστασία. Και οι δύο μηχανισμοί λειτουργούν συμπληρωματικά και ως ανταπόκριση σε κρίση αλλά και ως πρόληψη και προετοιμασία πριν από μια κρίση. Για τον έξους. Πρόκειται για κάτι που θεωρώ ότι είναι πολύτιμο και έχει ήδη αποδείξει την αξία του. Όταν πρόκειται για ε, το δίκτυο αυτό ανάμεσα στην ανθρωπιστική βοήθεια και την ανάπτυξη. Και θέλω να συνεχίσουμε με τον έξους. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί δεν θέλουμε η ανθρωπιστική βοήθεια να χρειάζεται για πάντα κάπου. Δεν μας εφέρει κάτι τέτοιο. Ούτε βέβαια συμφέρει τους δικαιούχους. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον τους, αλλά και προς το δικό μας συμφέρον, να βγουν από αυτή την κατάσταση εξάρτησης από την ανθρωπιστική βοήθεια. Και ακριβώς εδώ είναι που βλέπω και εγώ το ρόλο της ανάπτυξης. Εδώ έρχεται. Οπότε ανθρωπιστική βοήθεια και ανάπτυξη, νέξους. Εγώ θέλω την εμπλοκή του συναδέρφου ε, της κυρίας Ουρπιλάινεν που είναι για τις διεθνείς ε, σχέσεις και να υπάρχει αυτή η συνεργασία ήδη από την αρχή μεταξύ μας. Γιατί αν αντιμετωπίσετε τις πραγματικές αιτίες που οδηγούν σε μια ανθρωπιστική κρίση, βοηθάτε να περάσει κανείς από την ανθρωπιστική βοήθεια στην ανάπτυξη. Επίσης, το Nexus έχει επεκταθεί και έχει συμπεριλάβει και τη συνιστόσα της ειρήνης και έχει νόημα αυτό. Έχει νόημα γιατί υπάρχουν περιπτώσεις, Σομαλία για παράδειγμα, που δεν μπορούμε να έχουμε αναπτυξιακή συνεργασία όταν δεν υπάρχει ειρήνη. Οπότε πρέπει να πετύχουμε την ειρήνη στη Σομαλία αν θέλουμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη. Αν θέλουμε να βγάλουμε τον κόσμο από την εξάρτηση για αυτή. Ε, δεύτερη ερώτηση, παρακαλώ. Ο συνάδελφος Χόλβενι ανέφερε το παράδειγμα της Συρίας. Πιστεύω ότι εδώ είναι μεγάλη πρόκληση. Πώς φαντάζεστε τη συνεργασία με την Επίτροπο για την Ανάπτυξη και με την είπατε εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική και τον Αντιπρόεδρο Μπορέλ. Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να τονίσετε σε αυτούς τους οδητερούς αυτά που προωθούμε στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε ό,τι αφορά την Ατζέντα 2030. Οριστή Επίτροπος, παρακαλώ για απάντηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλευτά, για την συμπληρωματική αυτή ερώτηση. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συμμετέχω ε, σε αυτό το κομμάτι που θα αφορά τις εξωτερικές σχέσεις υπό αντιπρόεδρο για την πολιτική ασφάλειας. Νομίζω ότι είναι μια καλή λύση αυτή, γιατί δίχως άλλο η ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί μέρος της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως πρόκειται για κάτι πολύ ιδιαίτερο. Γιατί βασίζεται σε πολύ συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες είναι διαφορετικές από οτιδήποτε καθεντήριες γραμμές έχουμε για άλλου είδους εξωτερική δράση. Σκοπεύω λοιπόν να συνεργαστώ στενά με τους συναδέρφους σε, αυτό, αυτή την ομάδα εξωτερικής δράσης και να φροντίσω να τηρούνται οι ανθρωπιστικές αρχές. Ευχαριστούμε κύριος Γκέρενς. Κύριε Μελλοντική Επίτροπε, ανάμεσα στις αρχές τις ε, δράσεις της ανθρωπιστικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε και την αμεροληψία, που πιστεύω ότι είναι μία από τις πιο βασικές αρχές. Ε, ο ΙΕ, ε, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, η Εθνική Ερυθρή Σταυρή, οι διάφορες εθνικές ή διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν το τομέα είναι αμερόληπτες. Γιατί αυτός που χρειάζεται βοήθεια δεν μας ενδιαφέρει αν είναι με μας ή όχι. Δεν μπαίνουν τέτοια ερωτήματα. Το μόνο κριτήριο που οδηγεί σε ανθρωπιστική δράση είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κανείς ή οι λαοί που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Αν δεν τηρεί κανείς αυτή την αρχή, αυτό είναι μεγάλος κίνδυνος. Και γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ευρύ φάσμα ε, δυνατοτήτων παρέμβασης, μεταξύ άλλων την ανθρωπιστική βοήθεια. Οπότε επιτρέψτε μου να σας κάνω μία σύσταση ως Ευρωβουλευτής που έχει περάσει τέσσερις θητείες ανθρωπιστικής δράσης εδώ, σε αυτή την Επιτροπή, είναι να τηρήσετε με νύχια και δόντια αυτή την αρχή της αμεροληψίας. Γιατί αν δεχτεί επιθέσεις αυτή η αρχή, αν δεν τηρηθεί, αν κάποιος μπει στον πειρασμό να μην ανταποκριθεί σε αυτή την αρχή, τότε κινδυνεύει όχι μόνο η φήμη της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά εκτιθέμεθα σε κίνδυνο και όσοι δρούν επιτόπου εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Απάντηση, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμε κύριε Γκέρνες, και ευχαριστώ πολύ για την σύστασή σας. Δίνω ιδιαίτερη σημασία, γιατί έχετε τεράστια εμπειρία πράγματι. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Τώρα, θα ήθελα να πω τα εξή: Το να τηρεί κανείς αυτή την αρχή, δεν το βλέπω κάτι σαν κάτι δογματικό. Το να τηρεί κανείς αυτή την αρχή, όπως και την αρχή της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας, είναι μια αναγκαιότητα για να λειτουργήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να μας βλέπουν οι άλλοι σαν κάποιος που μεροληπτούν. Είμαστε δηλαδή σε μια εμπόλεμη σύγκρουση και είμαστε με τη μία με την άλλη πλευρά. Όχι. Αν αυτή ήταν η αντίληψη για μας, προφανώς και τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η ανθρωπιστική μας βοήθεια και η ανθρωπιστική μας ε, δράση. Δεν θα μας εμπιστευόταν ο κόσμος. Οι ίδιοι αυτοί που έχουν ανάγκη. Και πάνω απ' όλα βέβαια θα θέταμε σε κίνδυνο και τους ίδιους ε, τους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν επιτόπου την ανθρωπιστική βοήθεια. Φυσικά και το συνειδητοποιώ και είναι συνεκβάν μου αυτή η προϋπόθεση για την ανθρωπιστική βοήθεια, ιδιαιτερότητα και μεροληψία. Ωραία. Συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ. Η ερώτησή μου συμπληρωματική απαντήθηκε, δεν χρειάζεται να την ξαναθέσω. Ευχαριστώ κύριε Γκέρενς. Οικονομήσαμε και χρόνο. Μισελ Ριβαζή για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε υποψήφια επίτροπε. Νομίζω ότι απέχει η δική μου ερώτηση από αυτή του προηγουλαλήσαντος. Είσαστε επίτροπος για διαχείριση των κρίσεων. Δεν υπάρχει πλέον η ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτή τη διατύπωση. Ποια είναι τα κριτήρια παρέμβασης σε μια ανθρωπιστική κρίση. Όταν έχουν φυσικές καταστροφές, όπως το κυκλώνα στις Μπαχάμες και επισητιστικά προβλήματα, είναι σαφές, ε, παρεμβαίνει η Ευρώπη όταν όλα έχουν καταστραφεί. Όταν είναι κάπως πιο λεπτές οι διαφορές, όπως αυτό που συνέβη στην Ελλάδα, μετά από τα μέτρα λιτότητας, Πώς έδρασε η Ευρώπη να της Ελλάδα, όταν δεν είχαν πλέον πρόσβαση στα φάρμακα οι άνθρωποι όταν οι γυναίκες δεν μπορούν πλέον να έχουν ε, θεραπεία του καρκίνου τους ή να πάνε να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Αυτά τα εντάσσετε στην ανθρωπιστική βοήθεια εσείς. Για μένα δηλαδή θέλω να δω σε ποιο επίπεδο βάζετε τον πύχη. Ποια είναι τα κριτήρια παρέμβασης όσον αφορά τα θέματα τα συγκεκριμένα. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ αξιότιμη κυρία Χρυβαζή Να πω κάτι για τον τίτλο του χαρτοφυλακίου του Επιτρόπου. πρόθεσή μας ήταν να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει ένα μέλος αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι υπεύθυνο για ανταπόκριση σε κατεπίγουσες ανάγκες, ανταπόκριση σε κρίσεις. Προφανώς η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ένα κομμάτι, κομμάτι της ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Ενώσης σε κατεπίγους ανάγκη. Αλλά είναι διακριτό τμήμα. Διέπεται από ξεχωριστές αρχές και θα επιμείνω από αυτού. Η ερώτησή σας τώρα. Είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας. Ένα ερώτημα για όλους μας. Η απάντησή μου είναι εξή. Πρώτα απ' όλα κινούμεθα βάσει της αξιολόγησης αναγκών. Όταν αξιολογήσουμε ότι φύσταται ανάγκη πρέπει να πάμε. Σύμφωνα με την αρχή της αμεροληψίας. Και αν η ανάγκη υπάρχει εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει να κινηθούμε. Εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να στερήσουμε ανθρωπιστική βοήθεια από πληγέντες πληθυσμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για κάποια ενιολογική λόγο. Θα αντέβαινε τις αρχές που προανέφερα επανειλημμένα. Καταρχήν η απάντησή μου είναι καταφατική. Ναι, ναι. Ή αναγκαίων θα πρέπει να παρεμβαίνουμε και να κάνουμε ανθρωπιστικό έργο και εντός της Ένωσης. Συνέβη ήδη μια φορά μάλιστα. Με την κρίση τη μεταναστευτική Ανθρωπιστική βοήθεια χορηγήθηκε εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Στην Ελλάδα, για να βοηθήσουμε την Ελλάδα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, την πρόκληση αυτή. Ευχαριστώ. Διευκρινιστική ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση που συνδέεται με αυτή. Ας πούμε σεισμό στην ΑΕΤ. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, πώς συσχετίζουμε την κατάσταση, την κατεπίγουσα ανάγκη και την Απεμπλοκή από την κατάσταση. Όταν δώσαμε τρόφιμα στην Αιτή δεν ήταν για τον πληθυσμό. Θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, αυτό που τρώνε οι άνθρωποι. Μετά, οι σπόροι. Πολύ συχνά δώσαμε σπόρους, γενετικά τροποποιημένους συχνά σπόρους, που διατάραξαν τη γεωργία εν συνεχεία στον τόπο αυτό. Ποια στρατηγική θα εφαρμόσετε ούτω ώστε να συσχετίζεται η ανθρωπιστική βοήθεια με την αναπτυξιακή βοήθεια, να υπάρχει μια συνοχή. Διότι οι κατεπίγουσες αυτές παρεμβάσεις έχουν και συνέπειε εν συνεχεία. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, απάντηση πράγματι είναι ένα πρόβλημα πρόκληση για πολλού λόγους. Μεταξύ άλλων λόγων, επειδή οι διαδικασίε που ακολουθούμε για ανθρωπιστική βοήθεια είναι πιο ευέλικτες διότι πρέπει να δράσουμε γρήγορα, τάχιστα, για να σώσουμε ζωές και να μειώσουμε τα δεινά του πληθυσμού και έχουμε και τη διαδικασία για χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας, απ' την άλλη. Αυτές οι προκλήσεις μπορούν να υπερκεραστούν μέσω καλής συνεργασίας και θα συνεργαστώ, αυτή είναι η πρόθεσή μου, θα συνεργαστώ πολύ καλά με τον συνάδελφο Ούρτι Λάινεν, τη συνάδελφο Ούρτι Λάινεν, τα συζητήσαμε αυτά μαζί της συμφωνεί ότι πρέπει να το επεξεργαστούμε. Όσο πιο γρήγορα αυτοί οι δύο άξονες εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ενώσεως συνεργαστούν, το καλύτερο, τόσο το καλύτερο. Ευχαριστώ. Μπερνάρτ Σμινιόκ για το IT. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να χορηγήσουμε βοήθεια όπου αυτή χρειάζεται στον κόσμο. Αλλά πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να πάμε και πολύ μακριά, γιατί μπροστά στην πόρτα μας, στα εξωτερικά μας σύνορα, έχουμε μια πραγματική κρίση, μια κρίση η οποία ε, προκαλείται από ένα συνεχές, μια συνεχή ροή μεταναστών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι παράνομες δραστηριότητε που έμεσα ή άμεσα αποτελούν απειλή για τους πολίτες μας στην Ευρώπη, ή που υπονομεύουν τα οικονομικά συμφέροντα των κρατών μελών θα πρέπει να αποτραπούν, να περιοριστούν, να ανασταλούν. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου οι παράνομες ροές μεταναστών να σταματήσουν με βιώσιμο τρόπο, όπως λέμε στη μοντέρνα γλώσσα. Θα πρέπει τα εγκληματικά μοντέλα των ε, λάθρο, λαθεμπόρων ανθρώπων, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από τρίτες χώρες ή όχι, ή από κράτος μέλος ή οποιαδήποτε μικείο, να σταματήσουν άμεσα και για πάντα. Τι συγκεκριμένα λοιπόν μέτρα σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε προς την κατεύθυνση αυτή προκειμένου να περιοριστεί η παράνομη μετανάστευση στα εξωτερικά σύνορά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο υποψήφιος επιτροπός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ζημνιόκ. Θα ήθελα να τονίσω καταρχάς το εξής. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι ένα εργαλείο διαχείρισης μετανάστευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άλλα εργαλεία για το θέμα αυτό. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν συγκαταλέγεται σε αυτά. Κατά δεύτερον, όταν αξιολογούμε το κατά πόσο συντρέχει λόγος ανθρωπιστικής βοήθειας, συνήθως επικεντρωνόμαστε στα άτομα τα οποία εκτοπίζονται α, καταναγκαστικά πρόσφυγες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρνηθούμε την ανθρωπιστική βοήθεια σε μετανάστες, σε οικονομικούς μετανάστες για παράδειγμα. Όλος χερός, όπως είπα, όμως προηγουμένως έχουμε άλλα εργαλεία προς την κατεύθυνση αυτή. Αν υπάρχει όμως και ανθρωπιστική ανάγκη, ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, θα τη χορηγήσουμε και εκεί. Αυτό το κάνουμε για παράδειγμα στη Βοσνία, στη Βοσνία Ρισεκοβίνη, η οποία δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχεται. Παρά το γεγονός ότι τμήμα, ότι τμήμα των μεταναστών είναι ξεκάθαρα άνθρωποι οι οποίοι είναι οικονομικά μετανάστε, οικονομικοί μετανάστε. Δεν είναι πρόσφυγε, είναι μεικτέ οι μεταναστευτικέ ροέ όπω τι αποκαλούμε. Χορηγούμε ωστόσο ανθρωπιστική βοήθεια βάσει της ανάγκης που συντρέχει και όχι του στάτους ε, των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Η συμπληρωματική ερώτηση. Σημείωσα αυτά που μας είπατε, αλλά διαπιστώνω ότι ακόμα δραστηριοποιήσαστε και στις, δράσεις αντιμετώπισης κρίσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι κρίσεις αυτές δεν μπορούν να περιοριστούν στο ξέσπασμα ενός ηφαιστείου. Σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε τους πολίτες της Ευρώπης. Γιατί στην Ευρώπη δεν καταφέραμε πάντα να προστατεύσουμε τα σύνορά μα. Έχουμε τρομοκράτε με τρομοκρατικές ενέργειες, λάθρο εισαγωγέ ε, όπλων και ε, δεν θα ήθελα να έχουμε τέτοιες ε, μεγάλες απειλέ, οι οποίε και αυτέ αποτελούν κρίση για να προστατεύσουμε του πολίτε μα λοιπόν, του δικού μα πολίτε. Στην εντολή σας λοιπόν, στο χαρτοφυλόκιά σας, θα έχετε σίγουρα να εξετάσετε τέτοιες υποθέσεις. Το θέμα λοιπόν της διαφύλαξης των εξωτερικών συνορών έχει να κάνει και με αυτές τις ε, απειλές. Πώς θα προστατεύσετε τους πολίτες από ασθένειες, ε, για παράδειγμα, οι οποίες διαδίδονται, γιατί αυτοί οι άνθρωποι φέρνουν ασθένειες ε, οι παράνομοι μετανάστες, οι πρόσφυγες και πώς θέλετε να διατηρήσετε σε πιο προορισμένο βαθμό τέτοιες ε, περιπτώσεις μόλυνσης των πολιτών μας όπως ο έμπολα. Αυτό που από το και αν είναι εσείς. Ε, εμείς σκεφτόμαστε τους πολίτες της Ευρώπης. Γι' αυτό είστε εδώ, γι' αυτό πληρώνεστε. Όχι για να βελτιώσετε, να βελτιώσετε κάτι τον κόσμο ολόκληρο. Σας παρακαλώ λέει ο Πρόεδρος Εντάξει, Θα ήθελα, έχετε όλοι ένα λεπτό στη διάθεσή σας να υπενθυμίσω στα υπόλοιπα μέλη ότι θα έχουν την ευκαιρία, μάλλον κάθε μέλο έχει το δικαίωμα να θέσει την ερώτησή του. Να δώσουμε το λόγο στον υποψήφιο επίτροπο να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ και να πω ότι δεν έχουμε μεταναστευτική κρίση. Υπήρξε μεταναστευτική κρίση το 2015-2016. Τώρα, σε σχέση με την περίοδο εκείνη, τα πράγματα είναι λίγο πολύ έλεγχο. Ναι, Βεβαίως υπάρχουν μεταναστευτικές ροές, κάποιοι άνθρωποι από αυτούς χρειάζονται και ανθρωπιστική παγκόσμια μάλλον υποστήριξη και προστασία. Κάποιοι απλά θέλουν μια καλύτερη ζωή, το οποίο είναι ένα στόχος, ένας, μια επιθυμία ευσεβής. Θεωρώ όμως ότι η κατάσταση πλέον είναι λίγο πολύ υποέλεγχο και γι' αυτό λοιπόν ο Επίτροπος Ιστορικών Υποθέσεων θα αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά και ως μελλοντικό συντονιστής για θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια ανταπόκριση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κοψίνσκα τώρα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια η ανθρωπιστική κοινότητα έχει πάει προς τον ιδιωτικό τομέα. Γίνονται, υπάρχουν διάφορες συνεργασίες με διάφορες οργανώσεις και προσφέρονται μάλιστα και τεχνολογικές λύσεις προς συνεργασία. Τώρα, ο οριστής επίτροπος αναφέρθηκε και σε άλλους τομείς, αναφέρθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Ρωτάω λοιπόν εσείς τι πιστεύετε για το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην ανθρωπιστική βοήθεια. Θα ενισχύσετε το ρόλο του ιδιωτικού τομέα. Πέρα από τα όσα θεωρούμε δηλαδή σήμερα παραδοσιακά ως ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση αυτή. Όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν κενά, το 44% της, των αναγκών για ανθρωπιστική βοήθεια δεν καλύπτονται σήμερα. Οπότε φυσικά και θα έπρεπε να κοιτάξουμε τη δυνατότητα συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Τώρα, ένα πράγμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Ότι αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται σε βάρος των αρχών μας που διέπουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεύτερον, κανείς δεν πρέπει να είναι σε θέση να κάνει business από την ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτό πρέπει να σημειωθεί. Δεν πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο ποτέ. Δεν είναι επιλογή, δεν μας παίρνει για κάτι τέτοιο. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ε, ένας ευγενής σκοπός, ε, δεν είναι εμπορικός και ποτέ δεν πρέπει να καταστεί εμπορικός. Τώρα, βλέπω τη δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Εξάλλου πρόσφατα διαπιστώσαμε με τη σημερινή Επιτροπή. Είδαμε κάποια επέκταση σε πιο καινοτόμες προσεγγίσεις όπως μεταφορά ρευστού υπό την ε, μορφή χρεωστικών καρτών. Ο ιδιωτικός τομέας, ο τραπεζικός δεν χρεώνει με κόστος όπως κάνει συνήθως για να προσφερθεί αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν βγάζει κέρδος δηλαδή από αυτή τη μεταφορά χρημάτων. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και ισχύει σε διάφορους καταβλισμούς προσφύγων όπου ιδιωτικές εταιρείες βοηθούν είτε με ε, φωτοβολταϊκά. Είναι και αυτό κάτι που μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας. Αλλά επιμένω, όχι εμποριοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Όχι. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ και συμφωνώ, συμφωνώ με όσα είπατε. Κάνατε διάφορες προτάσεις, οπότε δεν έχω παρετέρω ερώτηση. Καλύπτομαι. Μιγέλ Κανκρέσπο, παρακαλώ. Ο κύριο Σουρμπάν Κρέσπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και εσά. Το πρώτο που θέλω να σχολιάσω είναι ε, το εξή, ότι δεν πρέπει να ακούμε πυροτεχνήματα. Δεύτερον, να ξέρετε ότι μας εξέπληξε πάρα πολύ που όπως είπε και συνάδελφος πριν από λίγο, το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας που δεν υπάρχει στο χαρτοφυλάκιο και δεν έχει εκπλήξει μόνο εμάς αλλά και την κοινωνία των πολιτών και όχι μόνο μας εκπλήσει αλλά και μας ανησυχεί επειδή είπατε εσείς ότι δεν είναι η ανθρωπιστική βοήθεια ε, μόνο ένα μέσο αντιμετώπισης και διαχείρισης μάλλον κρίσης. Δηλαδή η ανθρωπιστική βοήθεια βγαίνει τελικά από το χαρτοφυλάκιο. Ελπίζω όχι, βγήκε μόνο από τον τίτλο. Πάντως σας άκουσα όταν είπατε ότι μία από τις προτεραιότητές σας είναι το ανθρωπιστικό δίκαιο και η προστασία του. Γιατί ετίθεται σε κίνδυνο σε πολλά μέρη του κόσμου. Αφού είναι η προτεραιότητά σας λοιπόν, τι θα κάνετε κατά τη διάρκεια της θητείας σας ώστε να προστατεύσετε ακριβώς αυτό το δικαίωμα τι θα κάνετε. Ε, θα προτείνετε διακοπή εμπορικών συμφωνιών, αν ε, υπάρχει τέτοια παραβίαση. Θα επιβάλλετε κυρώσεις σε όσους δεν τηρούν αυτό το ανθρωπιστικό δίκαιο. Απάντηση. Ευχαριστώ για αυτήν την ε, ερώτησή σας. Νομίζω ότι είπα στην αρχή, στην παρουσίασή μου, πόσο μεγάλη σημασία έχει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και υπάρχουν παραβιάσεις όλο και περισσότερο. Και βλέπουμε πως επίτηδες γίνονται επιθέσεις ε, απέναντι σε ανθρωπιστικές υποδομές. Εμποδίζεται η πρόσβαση ε, του πληθυσμού που έχει ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια, εμποδίζεται η πρόσβασή τους αυτή. Τι θα κάνω, ναι, θα υψώσω τη φωνή μου, ναι. Θα καταδικάσω κάθε παραβίαση του ανθρωπιστικού διεθνούς δικαίου. Θα το κάνω. Δεύτερον, σκοπεύω να συνεργαστώ με τις οργανώσεις εκείνες που έχουν προνομιακή πρόσβαση σε κλάδους ε, με στρατό, είτε πρόκειται για κρατικό είτε όχι. Και θα επιμείνω στο πόσο μεγάλη σημασία έχει ο σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Υπάρχουν ε, τέτοιες οργανώσεις που έχουν προνομιακή πρόσβαση σε τέτοια στρατεύματα. Ο Ερθρός Σταυρός, για παράδειγμα. Οπότε βασίζομαι ότι θα έχω συνεργασία με αυτούς, ώστε σε κάθε περίπτωση σύγκρουσης να φροντίσουν να υπάρξει καλύτερο σεβασμός και προστασία βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Το άλλο που σκοπεύω να κάνω, το τρίτο, είναι το εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωρίζετε, έχει κάποιες αποστολές κατάρτισης ε, σε στρατιωτικές αποστολές για την ασφάλεια κλπ. Θα φροντίσω λοιπόν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση να συμπεριλάβουν στην κατάρτισή τους και θέματα όπως είναι ο σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, θέματα που έχουν να κάνουν με την ισότητα του φύλου κλπ. Ε, παρακαλώ, πληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Μα υπάρχει ένα πρόβλημα. Εδώ είμαστε ε, συνηθισμένοι να τα βάζουμε με την αδικία, με τις παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου. Εντάξει, αλλά θέλω κάτι συγκεκριμένο, οπότε σας κάνω τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις για τρία συγκεκριμένα πράγματα και σας ρωτώ τι θα κάνετε. Πρώτον, είπατε ότι, ότι γίνονται επιθέσεις σε ανθρωπιστικούς στόχους, όπως για παράδειγμα κάνει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Τι θα κάνετε λοιπόν και τι θα κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις που όντω υπάρχει κατάφορη επίθεση από πλευρά του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Δεύτερο, στην περίπτωση της Τουρκίας με τους Κούρδους. Τι θα κάνετε ή για την περίπτωση του Μαρόκου με, τις, ε, με τη Σαχέλ τι θα κάνετε. Είναι τρεις περιπτώσεις, τρία παραδείγματα παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου. Εμείς τα λέμε, αλλά δεν βλέπουμε να έρχεται κανένα, ε, κανένα αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, Σαουδική Αραβία με Ιεμένη. Τι έγινε, υπήρξε εμπάργο όπλων. Όχι. Τι θα κάνετε λοιπόν εσείς. Ευχαριστώ. Η απάντηση. Ναι, θα φωνάξω θα υψώσω τη φωνή μου, θα το κάνω δημόσια, αλλά επίσης θα χρησιμοποιήσω και ό,τι διόδους έχουμε στη διάθεσή μας, διακριτικά, άτυπα, μέσω οργανώσεων, όπως το είπα και πριν, προκειμένου να πείσω, να πείσω όλους τους φορείς. Ένοπλους στην περίπτωση ένοπλων συγκρούσεων για να σέβονται το ανθρωπιστικό δίκαιο δεν έχω αρμοδιότητα εξεταστική. Οπότε δεν μπορώ να βγω και να πω ότι με πρόθεση έγινε η παραβίαση αυτή, όπως υποψιαζόμαστε ότι ισχύει στην Συρία, όπου υπήρξαν επιθέσεις επίτηδες, ε, πιστεύω, ή να πω ότι ήταν κατά λάθο, όπως μπορεί να συμβαίνει αλλού. Χωρίς λοιπόν ξεκάθαρες απαντήσεις από αυτού, εγώ θα περιοριστώ να ε, καταγγείλω τις παραβιάσεις δημόσια και να χρησιμοποιήσω όλες τις διόδους που έχουμε στη διάθεσή μας, επίσημες και ανεπίσημες, για να πείσω να υπάρχει σεβασμός στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ευχαριστώ. Τελείωσε ο πρώτος γύρος με εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Τώρα θα μιλήσουν τα άλλα μέλη. Θα δώσω το λόγο στη Χίντεργαρτ Μπέντελε από το ΕΛΚ. Αξιότιμη κυρία υποψήφια Επίτροπε Ενέργεια, θα ήθελα να σας αναφέρω κάτι από τις πολιτικές ε, ε, τρει γραμμές της Ρωσόφαν Λάιεν. Η Ευρώπη έχει την ευθύνη να βοηθήσει τις χώρες και να παρέχει αξιοπρεπείς ε, ανθρωπιστικές συνθήκες. Υποστηρίζω λοιπόν τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων, τέλο παράθεση. Ε, Πώ λοιπόν τοποθετήσετε σε ό,τι αφορά την ιδέα τέτοιων ανθρωπιστικών διαδρόμων και πού θα δημιουργούσατε τετοιου διαδρομου σα ευχαριστώ, ο επιτροπο Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Δεν είμαι σε θέση νομίζω να ερμηνεύσω. Τα είπε η εκλεγής πρόεδρος και τι έχει υπόψη της. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όχι διάδρομο ανθρωπιστικό, πώς να το πω. Ανθρωπιστικά κινήματα. Ξέρετε ποια κατάσταση επικρατεί όπως τώρα. Σε κάποια από τα ελληνικά νησιά επικρατεί η κατάσταση αυτή. Όλα τα ελληνικά νησιά που είναι κοντά στις τουρκικές ακτές ε, έχουν φορτωθεί, κατακλειστεί από μετανάστες. Αυτό που χρειαζόμαστε εκεί και αυτό που κάνουν οι ελληνικές αρχές ήδη είναι να εξασφαλίζουμε ότι αυτή η κατάσταση θα διορθωθεί. Αν δεν μπορεί να κατασκευάσεις περισσότερα κτίρια και δυναμικότητα στα νησιά, θα πρέπει να μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι ε, στην υπηρετική χώρα. Δεν μπορεί να τους κρατάς σε τέτοιες συνθήκες. Είδαμε τι συνέβη. Είχαμε και τραγική απώλεια ζωής. Μια μητέρα και μια κόρη χάθηκαν, έχασαν τη ζωή τους. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε αυτά να συμβαίνουν στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να συμφιλειωθούμε με τέτοια γεγονότα. Να συμβαίνουν αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έπρεπε να συμβαίνουν. Υπάρχουν και άλλες καταστάσεις όπου χρειάζονται ανθρωπιστική διάδρομη. Σε περίπτωση ενόπλων σειράξεων Πρέπει να εκενωθούν οι άμαχοι για να αποφύγει κανείς θύματα ή επιδείνωση ανθρωπιστικής κρίσης. Εκεί χρειάζονται ανθρωπιστικοί διάδρομοι για τους μη μάχημους, για τους άμαχους, για να οι άμαχοι να μεταφέρονται σε ασφαλή τοποθεσία. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας. σε ό,τι αφορά την ερμηνεία α, της κυρίας Φαντερ Λάιν αυτών που δήλωσε, κινηθείτε λίγο πιο μακριά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικό το θέμα αυτό για μας και νομίζω ότι και το θέμα α, του ανθρωπιστικών διαδρόμων έχει να κάνει με την ίδρυση τέτοιων διαδρόμων εκεί που υπάρχουν οι κρίσεις. Πού, λοιπόν, επί που σε περιπτώσεις κρίσεων μπορείτε να φανταστείτε ότι ενδεχομένω θα υπάρξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι τους επόμενου μήνε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε. μπορώ εύκολα να φανταστώ πολλά σημεία, πολλά μέρη, όπου ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν αναγκαίο. Η εμένη είναι μια περίσταση. Εκεί έχουμε τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση πιθανότατα αυτή τη στιγμή. Με το μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. 20 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ιεμένη και έχουμε και πόλεμο ταυτόχρονα. Έναν πολύ άγριο πόλεμο. Ναι, θα έπρεπε να υπάρχει μια δυνατότητα, ένα τρόπο να προστατεύσει κανεί του άμαχου, του πολίτε, κυρίω ευάλωτε ομάδε. Και να μετακινηθούν οι άμαχοι σε ασφαλέστερε περιοχέ. Εκτό των περιοχών των συγκρούσεων. Σας ευχαριστώ. Μόνικα Σιλβάνα Γκονζάλες, Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κλιματική αλλαγή. Κανείς δεν την αρνείται. Αναφερθήκατε και εσείς στην αρχική σας παρουσίαση και όλοι οι εμπειρογνώμονες λένε ότι περίπου 500 εκατομμύρια άνθρωποι, φανταστείτε ολόκληρη δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στα επόμενα 50 χρόνια θα αναγκαστούν να εκτοπιστούν Ασία, Μπαγκλαντές και αλλού, αλλά και Λατινική Αμερική, Αφρική και αλλού. Η κλιματική ε, αλλαγή θα θέσει σε κίνδυνο το νερό και την διατροφή ε, στην Ευρώπη. Και έχουμε και την μετανάστευση για ε, λόγους κλιματικής αλλαγής. Έχουν όμως ανθρώπινο πρόσωπο. Τι θα κάνουμε με αυτούς. Η κρίση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και Χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά φεύγουν και αφήνουν τα σπίτια τους για να σωθούν. Όμως η απάντηση, η διεθνής και η ευρωπαϊκή, ήταν περιορισμένη. Οπότε εσείς, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι θα κάνετε για δεδομένου ότι δεν υπάρχει επίσημο καθεστώς για αυτούς τους κλιματικούς πρόσφυγες. Κύριε Υποψήφη Επίτροπε, ευχαριστώ, αξιότιμο μέλος, για αυτή την άκρος επίκαιρη ερώτηση. Πάρα πολύ επίκαιρο θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα και ταχύτερα. Όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τον αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος. Κάτι που ήδη αισθανόμαστε. Αναφέρατε κάποιες περιοχές στην Αφρική. Ναι, το Σαχέλ και το κέρας της Αφρικής είναι οι περιοχές που ήδη γίνεται πολύ αισθητό ο αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος. Και υπάρχουν ήδη μετακινήσεις εκατομμυρίων ανθρώπων που λόγω της αλλαγής του κλίματος, του αντικτύπου της αλλαγής του κλίματος μετακινούνται. Εγώ θα δίσταζα παρόλα αυτά να τους αποκαλέσω αυτούς τους ανθρώπους σαν ε, κλιματικούς πρόσφυγες. Τη λέξη πρόσφυγας ίσως θα έπρεπε να αφήσουμε να καλύπτει πολύ ακριβή κατηγορία ανθρώπων που καθορίζεται πολύ ακριβώς στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς των προσφύγων. Άλλοι τους αποκαλούν εκτοπισθέντες λόγω κλιματικής αλλαγής, γιατί μπορεί να εκτοπιστούν εντός των χωρών τους. Ο ορισμός του ΟΗΕ για πρόσφυγα είναι κάποιος που ε, έφυγε από τη χώρα του ή χώρα της. Οι περισσότεροι από αυτούς που εκτοπίζονται λόγω αλλαγής του κλίματος μετακινούνται εντός της χώρας τους και πρέπει να βοηθήσουμε και αυτούς. Ε, πώς? Το ένα είναι πρόληψη. Προτίθεμαι να συνεργαστώ στενά με τον εκτελεστικό την που είναι υπεύθυνο για την Πράσινη Συμφωνία, το Ευρωπαϊκό Green Deal. Πρέπει να κάνουμε εδώ, να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μα στην Ευρώπη, να μειώσουμε τι εκπομπέ. Και το κλιματικό μας ίχνος. Μετά πρέπει να συνεργαστούμε με άλλε χώρε του κόσμου για να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Αυτό που δεν μπορούμε να αποφύγουμε πλέον όμω, ε, πρέπει να το, να το διορθώσουμε μέσω προσαρμογής. Ε, συμπληρωματική ερώτηση. Ε, ναι. Ακριβώς εκεί είναι το πρόβλημα, ότι οι προβλέψεις είναι πολύ ανησυχητικές και η προστασία των ανθρώπων αυτών που εσείς δεν θέλετε να τους ονομάζουμε κλιματικούς πρόσφυγες, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα, ότι αν τους ονομάσουμε κλιματικούς πρόσφυγες μπορούμε να τους προστατεύσουμε. Οι άνθρωποι αυτοί δεν καλύπτονται. Η σύμβαση του 51 της Γενέβης δεν τους συμπεριλαμβάνει όπως είπατε και εσείς. Οπότε γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε και η Ευρώπη να ηγηθεί και να συμφωνήσει και ο υπόλοιπος κόσμος μετά, ώστε να υπάρξει ένα καθεστώς για αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε, προβλέπετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσετε και να μην τους ονομάζετε απλώς κλιματικά εκτοπισμένους, αλλά να βρείτε και κάτι άλλο για να αποφύγουμε και τα διάφορα ξενοφοβικά που ακούσαμε ακόμα και σήμερα το απόγευμα εδώ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, ευχαριστώ Ακούω όλα τα σχόλια βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με όλα αυτά που ακούω. Αντιθέτως, υπήρξαν κάποια με τα οποία σαφώς διαφωνώ. Δεσμεύομαι να συνεργαστώ κυρίως με τον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ είναι θεματοφύλακας της συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς των προσφύγων. Θα συνεργαστώ με τους εταίρους μας. Όσον αφορά τον ορισμό του φαινομένου που περιγράψατε. Διότι υπάρχει κάτι σαφέ. Αυτοί οι άνθρωποι χρήζουν προστασία. Πρέπει να επεξεργαστούμε το θέμα της πρόληψης και της προσαρμογής στο κλίμα. Αν δεν κάνουμε τίποτα θα έχουμε εκατομμύρια, εκατομμύρια ανθρώπους που θα μετακινούνται. Πρέπει να προλάβουμε, να προσαρμοστούμε, να βοηθήσουμε να προσαρμοστούν. Δεσμεύομαι να συνεργαστώ με τους εταίρους του συστήματος του ΟΗΕ κυρίως για να πετύχουμε έναν καλό εφαρμόσιμο ορισμό για αυτούς τους ανθρώπους που σαφώς χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι βοήθεια. Χρυσούλα Ζαχαρόπουλου για το Ρινιού. Οι γυναίκες και τα κορίτσια σε περίπτωση συγκρούσεων είναι ε, πιο... τα θύματα τα οποία κινδυνεύουν περισσότερο. Πρόκειται για εγκλήματα, σεξουαλικά και άλλα, τα οποία επαναλαμβάνονται και μάλιστα τη μορυτή. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δρά στην ε, ανθρωπιστική βοήθεια, πρέπει επιγόντως να βρει μια λύση για αυτό το πρόβλημα. Στις γραπτές σας απαντήσεις λέτε ότι θα προωθήσετε την πρόληψη των σεξουαλικών αυτών βιωτήτων. Στην πράξη τι θα κάνετε ακριβώς και πώς θα συνεισφέρετε στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια μέσα από το δικό σας χαρτοφυλάκιο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, οριστής Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να φανταστώ ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς χωρίς να αντιμετωπίσουμε τις ειδικέ ανάγκες των πιο ευάλωτων ομάδων, κυρίως των γυναικών και των κοριτσιών. Στο δικό μας ανθρωπιστικό έργο, προφανώς οι γυναίκες και τα κορίτσια εκτίθενται στον κίνδυνο βίας σε βάρος των γυναικών κοριτσιών και συχνά, πολύ συχνά είναι και θύματα τέτοιων βιωτήτων. Γι' αυτό και πρέπει η ανθρωπιστική βοήθεια να λαμβάνει υπόψη αυτές τις περιπτώσεις και πρέπει να συμπεριλαμβάνει μέτρα σε όλα τα στάδια της ανθρωπιστικής μας βοήθειας. Πρόληψη, προστασία, με απλά μέτρα μπορεί να είναι πολύ απλά. Ας πούμε σε έναν καταβλισμό προσφύγων μπορούμε να κάνουμε πολλά για την ασφάλεια και την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών, βάζοντας χωριστές τουαλέτες με φώτα και με κλειδαριές. Κάτι το οποίο οδηγεί σε μείωση του κινδύνου ε, βίας σεξουαλική σε βάρος τους. Αυτή είναι μία λύση. Αλλά βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτές τις ειδικές ανάγκες και αυτές οι ειδικές ανάγκες συμπεριλαμβάνουν και την σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία. Πάντα όταν έχουμε να κάνουμε με θύματα βία σε βάρος ε, γυναικών. Συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κινδυνεύει και η εκπαίδευση. Και πάλι είναι τα κορίτσια που κινδυνεύουν περισσότερο και κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο, κάτι το οποίο τους εκθέτει ακόμα περισσότερο στη βία και στην σεξουαλική εκμετάλλευση. Όμως η εκπαίδευση δεν αποτελεί προτεραιότητα όταν πρόκειται για τους πόρους ανθρωπιστικής βοήθειας. Οπότε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω εσείς πώς θα ενισχύσετε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλίσετε τη συνέχιση της εκπαίδευσης ε, για τα κορίτσια που είναι τα περισσότερο ευάλωτα θα φροντίσετε να υπάρξουν τα κατάλληλα κονδύλια. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, οριστής Επίτροπος. Σας ευχαριστώ για την δεύτερη αυτή ερώτησή σας. Η εκπαίδευση θα αποτελέσει μία από τις προτεραιότητές μου όταν θα φροντίζω για ανθρωπιστική βοήθεια. Παραδοσιακά, η ανθρωπιστική βοήθεια ήταν τρόφιμα, ε, στέγαση κλπ. Ξέρουμε όμως ότι όταν φτάνει ο Σεπτέμβριος τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο. Δεν μπορούν να περιμένουν, ε, δεν ξέρω εγώ τι ανθρωπιστική κατάσταση να λυθεί, να αρχίσει ανάπτυξη κλπ. κλπ. Όχι, πρέπει να πάνε στο σχολείο, να γραφτούν στα σχολιά. Και αυτό είναι κάτι που αφορά και κορίτσια και αγόρια. Δεν υπάρχει διάκριση όταν πρόκειται για την εκπαίδευση. Καμία διάκριση, απολύτως. Καθόλου. Αυτή είναι μια από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα επιμείνω να φροντίσουμε η εκπαίδευση να παρέχεται και να προσφέρονται αρκετά κονδύλια γι' αυτό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε γενιές να πηγαίνουν χαμένες, τα κορίτσια να μην πηγαίνουν ε, στο σχολείο επειδή υπάρχει κάποια εκτακτή κατάσταση. Όχι. Να φροντίσουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις να προσφέρετε εκπαίδευση στα παιδιά. Να δώσω το λόγο στη Ράσα Γιουγνεβιτσκένε από το ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω λιθουανικά. Η ρατιολογική και πρινική κίνδυνη και οι κατεπίγουσες καταστάσεις είναι ε, περιστατικά χαμηλής ε, πιθανότητας. Στο, στην επιστολή αποστολή σας είπατε ότι θέλετε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξοπλίσει το μηχανισμό Rescue. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν σωστή χρηματοδότηση προς τον μηχανισμό αυτό και να υπάρχει και σωστή στελέχωση για τέτοιες είδους, τέτοιου είδους κατεπίγουσες ανάγκες. Τι επίπεδο ετοιμότητα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοιου είδου απειλέ, ραδιολογικέ και πυρηνικέ απειλέ, Πώ σκοπεύετε να ενισχύσετε τα εξωτερικά μα σύνορα προ την κατεύθυνση αυτή, Πώ θα εξασφαλίσετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να αυξήσει την ασφάλεια παλιών πυρηνικών εγκαταστάσεων ε, στα σύνορά τη ανατολικά και στα νότια των συνόρων. Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί τέτοιο τμήμα στην εντολή σας. Ευχαριστώ πολύ η απάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή και πραγματικά είναι ένα από τα θέματα τα οποία συμπεριλήφθησαν στο, στην επιστολή αποστολή μου και προφανώς και θα τα πάρω όλα αυτά στα σοβαρά γιατί είναι μέλος της αποστολή μου. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δεν είναι προετοιμασμένη για τέτοια περιστατικά. Τα είπατε χαμηλής πιθανότητας αλλά μεγάλης, μεγάλο αντικτύπου. Έτσι τα αποκαλέσατε. Ακριβώ επειδή είναι χαμηλή η πιθανότητα να παρουσιαστούν τέτοια περιστατικά. Θυμάμαι καιρού όπου υπήρχαν ψηλέ πιθανότητε τέτοιων ε, πυρηνικών κρίσεων στο ψυχρό πόλεμο. Θυμάμαι στη δική μου χώρα. Κανένα κτίριο, μεγάλο κτίριο, ούτε καν εκκλησία δεν μπορούσε να οικοδομηθεί χωρί πυρηνικό καταφύγιο. Σήμερα θεωρούμε ότι αυτά πλέον είναι του παρελθόντος. Έχετε δίκιο όμως, όλα αυτά θα μπορούσαν να συμβούν και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι δύσκολο να κινητοποιήσουμε τα κρατημέλη να προετοιμαστούν για κάτι το οποίο είναι, εκτιμούμε, έχει χαμηλές πιθανότητες να παρουσιαστεί. Εδώ πιστεύω ότι είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τέτοια μέτρα προετοιμασία για τέτοια περιστατικά πυρηνικών κρίσεων, για παράδειγμα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να οργανωθεί καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ότι στα διάφορα κρατημέλη ξεχωριστά για πρέπει να λάβουμε υπόψη ενώ χρειάζεται χρηματοδότηση, η οποία φαντάζομαι είναι πολύ υψηλή για κάθε κρατο μελο ξεχωριστά. Κατά δεύτερον, ε, αντίκτυπος, ε, ε, ο αντικτυπο τέτοιων κρίσεων δεν γνωρίζει σύνορα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, ωστόσο, το γεγονο ότι η πολιτική προστασία είναι πρωταρχικά αρμοδιότητα των κρατών μελών και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει συμπληρωματικό μόνο, υποβοητικό μόνο ρόλο. Αλλά σκοπεύω να το εξετάσω αυτό σοβαρά και να συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη για να τα πείσω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, γιατί όταν συμβαίνει μια κρίση και δεν είμαστε προετοιμασμένοι, είναι πολύ αργά πλέον. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση. Θα συνεχίσω στα λιθουανικά. Σε ό,τι αφορά ένα συγκεκριμένο πυρηνικό εργοστάσιο στην Λευκορωσία. Το Αστραβιτς ε, στη Λευκορωσία λοιπόν είναι ένα πυρηνικό εργοστάσιο το οποίο αποτελεί άμεση απειλή για τους πολίτες ε, της Ευρώπης. 20 χιλιόμετρα μόνο μακριά από τα εξωτερικά σύνορα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά παράβαση των σχετικών προτύπων συχνά λαμβάνουμε αναφορές για περιστατικά στο εργοστάσιο αυτό. Πώς θα χορηγήσετε πρακτική βοήθεια στα κράτη-μέλη που πλήττονται. Συμφωνείτε με την ε, άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αναστολή ε, ε, βοήθεια στις χώρες αυτές αν υπάρχουν συστηματικές παραβιάσεις των πρότυπων ασφαλείας. Θα θέλαμε λοιπόν επιπλέον ε, χρηματοδότηση για να υπάρχει ασφάλεια. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να οικοδημούνται τέτοιε εγκαταστάσει ε, όσο πιο μακριά γίνεται και να πρέπει να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των ε, πολιτών που κατοικούν κοντά στο εργοστάσιο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα να κάνω εικασίε για το επίπεδο ασφάλεια οποιαδήποτε μεμονωμένη σε κατάσταση για παραγωγή ενέργεια. Πολλά μπορούν να συμβούν και τέτοια προστατικά παρουσιάζονται παντού. Στη Φοκουσίμα πριν από πρόσφατα σχετικά, παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία και η ασφάλεια της εγκατάστασης θεωρούνταν όχι μόνο υψηλή, αλλά συμβατεί με όλα τα πρότυπα IAA. Όλα λοιπόν αυτά μπορούν να συμβούν. Ναι λοιπόν, η απάντησή μου είναι ναι. Σκοπεύω να δουλέψω για να αναπτυχθεί το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση τέτοιων ε, περιστατικών χαμηλής πιθανότητας αλλά υψηλού αντικτύπου όπως είναι οι ραδιολογικές και πυρηνικές καταστροφές. Έχουν συμβεί αυτά στο παρελθόν. Το Τσέρνομπιλ έγινε, συνέβησε. Άρα, απαντώ καταφατικά. Μάλιστα, θα εργαστώ προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά εδώ θα ζητήσω και την κατανόησή σας. Θα πρέπει να έχω την υποστηρίξη των κρατών μελών η πολιτική προστασία πρωταρχικά είναι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά θα παλέψω για να πάρω την υποστήριξή τους. Ευχαριστώ. Ευήν Ευήνιν Σύρ για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να συνεχίσω στα Σουηδικά, αν μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε υποψήφιε Επίτροπε Λένατσιτς. Είναι χαρά για μένα που άκουσα να λέτε ότι θέλετε να υποστηρίξετε τις αρχές της ανθρωπιστικής βοηθείας και ότι δεν θα κάνετε συμβιβασμό επ' αυτών. Και έρχομαι στην ερώτησή μου. Το 2016, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής Διεθνούς, ξεκίνησε ένα παζάρι, ένα, μια συμφωνία συνήθι μεταξύ δωρητών και των διαφόρων φορέων που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια για να γίνει πιο αποτελεσματική χορήγηση βοήθεια. Ήταν μια πρωτοβουλία που υποστηρίχθηκε από πάνω από 50 οργανισμούς και φορείς και από χώρε. Πολλοί εταίροι και της Γενικής Διευθύνσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ανθρωπιστική Βοήθεια και για την προστασία των πολιτών συμμετείχαν. Και πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ήθαν συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ανθρωπιστική βοήθεια μέσω τριών πυλώνων του ΟΗΕ, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και του Ερυθρού Σταυρού. Η ΜΚΟ είναι σημαντική σαν εκτελεστική φορής για ανθρωπιστική βοήθεια επιτόπια. Η ερώτησή μου, εσείς πώς βλέπετε τις μη κρατικέ οργανώσεις, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τι ρόλο παίζουν όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια και πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εγγυηθεί ότι υπάρχει αρκετή ποικιλομορφία εταίρων στην εκτέλεση των αποστολών ανθρωπιστικής βοηθείας, βλέποντας τους περιορισμούς τους οικονομικούς που έχει. Κύριε Επίτροπε, υποψήφια Επίτροπε. Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Θυμάμαι τη Σύνοδο Κορυφή στην Κωνσταντινούπολη αυτή για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη μεγάλη συμφωνία, το Grand Bargain. Θα επιμείνω επιπιστής εφαρμογής όλων των υποχρεώσεων, των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως για το Grand Bargain. Μου είπαν συνάδελφοι από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να προεδρεύει, συμπροεδρεύει στην ομάδα εργασίας για την υλοποίηση της Μεγάλης Συμφωνίας του Grand Bargain. Ένα σημαντικό τμήμα αυτής της συμφωνίας σχετίζεται με τους εταίρους, τους συνεργάτες μας, τους διάφορους φορείς, μεταξύ αυτών και πολλές ΜΚΟ. Είναι έμπιστοι οι εταίροι μας. Ελπίζω ότι και οι δύο πλευρές θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν στο Grand Bargain. Απλούστευση της υποβολής των εκθέσεων και αναφορών. Θα ακολουθήσω αυτή την κατεύθυνση. Ακολουθώντας αυτή την κατεύθυνση ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί. Δεν πρέπει να υπονομεύσουμε τους αναγκαίους ελέγχους και διαβεβαιώσεις που πρέπει να υφίστανται για να εξασφαλίσουμε συνετή, ορθή οικονομική διαχείριση. Δεν θέλω να ξεσπάσει κάποιο άλλο σκάνδαλο στο μέλλον όπου ανθρωπιστική βοήθεια ε, παρεξέκλεινε ήταν αντικείμενο κακής διαχείρισης, ε, κάποια απάτη διαπιστώθηκε. Πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες των ΜΚΟ, απαιτώντας ταυτόχρονα τα σωστά ελεγκτικά μέτρα και διαβεβαιώσεις όσον αφορά την οικονομική διαχείριση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάτι άλλο για τις τοπικές ΜΚΟ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό το ανέφερα ήδη στην ομιλία μου, θα ενθαρρύνω τους εταίρους μας, που είναι πάνω από 200, θα ενθαρρύνω τους εταίρους μας να εμπλέξουν τοπικές μικιό για τους προαναφερθέντες λόγους. Τους εξήγησα στην παρέμβασή μου. Άλλη την συμπληρωματική ερώτηση. Και ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω στα Σουηδικά. Πρέπει να πω ότι σας ευχαριστώ για την πολύ καλή σας απάντηση. Απαντήσατε και στην άλλη ερώτηση που ήθελα να σας θέσω. Για τους τοπικούς εταίρους, τοπικούς φορείς είχα κάποια ερώτηση. Και πρέπει να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν και αυτοί οι φορείς. Ήδη υπενθυμίσατε πριν ότι γνωρίζουν καλύτερα αυτή το τοπικό πλαίσιο για τη δράση. Σας ευχαριστώ λοιπόν και για αυτές τις σκέψεις και σταματάω εδώ. Παρακαλώ να απαντήσει η follow Επιτροπός. Ευχαριστώ και για αυτή την ερώτηση. Πολλοί εταίροι με τους οποίους συνεργαζόμαστε ήδη εμπλέκουν και συνεργάζονται με τοπικούς φορείς, εθνικούς ε, οργανισμούς, ΜΚΙΟ εκπροσωπούνται όπως η Διεθνής Ομοσπονδία ε, του Ερυθρού Σταυρού και διάφοροι άλλοι φορείς έχουν ε, τοπικούς εκπροσώπους. Είναι μία από τις υποχρεώσεις και δεσμεύσει θα λάβω πολύ σοβαρά. Θα προωθήσω με συνέπεια τη συμπερίληψη και συμμετοχή των τοπικών φορέων και στις ανθρωπιστικές δραστηριότητες καθώς και στην αύξηση των δυνατοτήτων που θα έχουν να κινηθούν στον τομέα και να συμπεριλαμβάνονται και σε εθνικούς συντονιστικούς μηχανισμούς ώστε να συμμετέχουν πολύ ενεργά στον όλο κύκλο ανθρωπιστικής βοήθειας. Να δώσω το λόγο τώρα στον Έρικ Μάρκαρτ από τους Πράσινους. Σας ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση από το πίσω μέρος της αίθουσας μάλλον ε, από το Προεδρείο. Στα γερμανικά θα κάνω την ερωτήση μου. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι εδώ στην Ευρώπη που έχουμε πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, και σχεδόν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι που κάποιοι από εμάς είμαστε τόσο μακριά από τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου και έχετε χρόνο να φανταστείτε ότι ε, εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε σε χειρότερη θέση και πληττόμεθα από τα προβλήματα του κόσμου γιατί οι ΜΚΟ έχουν ε, καταλήξει στο συμπέρασμα και είναι λίγο κρίμα γιατί και εγώ την ίδια ερώτηση θέλω να κάνω. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να κοιτάξετε το εξής, να μας πείτε πώς οι μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να υποστηριχθούν με ακόμα καλύτερο τρόπο και πώς θα εξασφαλίσετε να έχουν πρόσβαση σε εσά οι άνθρωποι οι οποίοι επιτόπου ζουν την πραγματικότητα και πολλά έχουν να μας πούν για το πώς δουλεύουν επιτόπου. Πώς θα ε, αναλάβετε την ευθύνη σας αυτή. Ο υποψήφιος επιτροπός. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά οι μη κυβερνητικέ οργανώσει. είναι από τους πιο αξιόπιστους και πολύτιμους εταίρους μας. Δυσκολεύομαι να φανταστώ το πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε το ανθρωπιστικό μας έργο, να δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς τις... ΜΚΙΟ. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι το Grand Bargain αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία. Αν όλοι ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, για να έχουμε ακόμα καλύτερη συνεργασία. Αλλά αυτό σημαίνει ότι και από πλευρά μας θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια. Δεν θέλουμε, για παράδειγμα, να υπάρχει μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια, μεγάλο ποσοστό της ανθρωπιστικής βοήθειας να πηγαίνει σε αντικειτικές δράσεις. Με το Grand Bargain, λοιπόν, αυτό, αναλήφθηκε δέσμευση. Όλοι να εργαστούν προς την κατεύθυνση μείωσης αυτού του ποσοστού. Εδώ λοιπόν είναι ένα παράδειγμα για ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να συνεργαστούμε με τη ΣΜΚΙΟ. Κατά δεύτερον, ένα ιδιαίτερο σημείο σε ό,τι αφορά τις τοπικές και εθνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Συχνά έχουν προβλήματα ικανοτήτων για την κινητοποίηση, για παράδειγμα, πόρων για την ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην ετοιμότητα και στο συντονισμό. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αυξήσουμε τις ικανότητές τους, γιατί όσο πιο πολλά μπορούν να κάνουν, τόσο καλύτερο θα είναι αυτό για, τους, για τον κόσμο επιτόπου, για τον πληθυσμό που ζει επιτόπου. Και αυτό θα πρέπει να το προωθήσουμε από κάθε άποψη. Να μην έρχεται βοήθεια από μακριά, δηλαδή από ανθρώπους μακριά προς τους ντόπιου πληθυσμού. Θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά αν είναι κοντά στην πηγή. Ευχαριστώ πολύ και τώρα η συμπληρωματική ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση αυτή. Αναφέρατε επίσης ότι δεν είναι δυνατόν κάποιες ΜΚΟ να μην μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, να μην μπορούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί. Και παρατηρούμε λοιπόν το εξή. Και μάλιστα όχι πολύ μακριά από εμά, αλλά στα εξωτερικά μας σύνορα, ε, πολλοί ανθρωπιστικοί φορείς δεν ε, μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Χιλιάδες άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο το περασμένο έτος. Τι θα κάνετε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή, θα κάνετε να ακουστεί η φωνή σας για να υποστηριχθούν οι ΜΚΟ που σώζουν ανθρώπινες ζωές στη Μεσόγειο. Η απάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή, η οποία μου επιτρέπει να δηλώσω με πάσα σαφήνεια ότι είμαι πεπισμένος ότι η ανθρωπιστική δραστηριότητα ποτέ δεν θα πρέπει να υπόκειται σε, με εγκληματικές, σε εγκληματικές κυρώσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο και θα το επαναλάβω αυτό όσο συχνά χρειαστεί. Δεν είναι δυνατόν να διώκουμε κάποιον για την προσπάθεια που έκανε στον ανθρωπιστικό κλάδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εκ παραλληλού. Μιλήσατε για τη Μεσόγειο. Υπάρχουν κανόνες ό,τι αφορά τη θαλάσσια διάσωση. Οι κανόνες αυτοί δίνουν συγκεκριμένες ευθύνες στα κρατημέλη. θα πρέπει να τηρείτε το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο για την ανθρωπιστική βοήθεια, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά εφαρμόζονται λοιπόν. Ευχαριστούμε. Τώρα η κυρία Γιάννα Κάντσι έχει το λόγο. Παρακαλώ. Θα μιλήσω Ιταλικά. Πριν θέσω το ερώτημά μου στον υποψήφιο επίτροπο, θα ήθελα να εκφράσω κάτι. Στον ορισμό των στόχων και των αποτελεσμάτων που προσδοκούμε, πάντα είναι κανά να, να έχουμε και μια δόση ρεαλισμού όταν θέτουμε στόχους. Και γι' αυτό θα ήταν σημαντικό να έχουμε έναν ορισμό των προτεραιοτήτων που θα ακολουθήσουμε, έχοντας υπόψη τις πιο μεγάλες κρίσεις που πρέπει αντιμετωπιστούν και ποια είναι τα πλαίσια εντός των οποίων η παρέμβασή μας μπορεί ε, να δώσει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Από αυτή την οπτική γωνία λοιπόν, ξεκινώντας, κύριε Λέναρτσιτς, στην επιστολή σας ε, είπατε ότι θέλετε να εργαστείτε με του μελλοντικού ε, επιτρόπους για να κατέξετε πολιτικές που θα δώσουν ε, λύσει για ανθρωπιστικά θέματα, για ασφάλεια και ανάπτυξη. Θέλω να καταλάβω ποια εργαλεία θα θέλετε να υποστηρίξετε για να αντιμετωπίσετε τα αίτια που είναι η ρίζα της, των μαζικών μεταναστεύσεων που ενδιαφέρουν άμεσα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, απάντηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ανέφερα τις προτεραιότητές μου. Και ευχαρίστως να επεκταθώ περισσότερο. Εσείς αναφέρεστε σε μακροπρόθεσμες λύσεις. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι για άμεση ανακούφιση. Η ανθρωπιστική βοήθεια έχει ως στόχο ε, επίγουσες ανάγκες. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν και άλλα πιο μακροπρόθεσμα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Γιατί όπως είπα και νωρίτερα, πρέπει να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση του ντόπιου πληθυσμού για να φροντίσουμε να επιστρέψουν στην κανονικότητα. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε με την διασύνδεση αυτή της ανθρωπιστικής βοήθειας με την ανάπτυξη, με αυτή τη σύνδεση. Και συνεργάζομαι και θα συνεργάζομαι με την κυρία Φοντερ ώστε ευθύ εξ αρχής να έχουμε και αυτήν την μακροπρόθεσμη διάσταση κάθε φορά που αυτό καθίσταται δυνατό, ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και τις πιο μακροπρόθεσμες ανάγκες του ντόπιου πληθυσμού. Υπάρχει και μια άλλη σημαντική πτυχή που σκοπεύω να καλύψω και αυτή είναι η πρόληψη. Και η αντίσταση, η αντοχή ε, που μπορεί να αποκτήσει ο κόσμος πριν την επόμενη κρίση, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει καλύτερα την επόμενη κρίση. Και να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο μέρος των ανθρωπιστικών μας δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνουν και αυτήν την διάσταση, δηλαδή μείωση του κινδύνου, του υπερχόμενου κινδύνου. Δεύτερη ερώτηση. Συμπληρωματική ερώτηση. Όχι, καλώς. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, συνεχίζουμε. Γιάννα Κοψίνσκα. Ευχαριστώ πολύ. Τα τελευταία χρόνια οι φυσικές καταστροφές έπληξαν σχεδόν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, προκάλεσαν πολλούς θανάτους, τραυματισμούς και εκατομμύρια σε ζημιές, σε υποδομές. Είχαμε πλημμύρες, πολλές καταστροφές που δοκίμασαν το σύστημα αντίδρασης αντιμετώπιση των κρίσεων των κρατών μελών. Δηλαδή έφτασε αυτά τα συστήματα στα όρια τους. Φόβοι περί ασφαλείας επίσης είναι πιο περίπλοκοι, πιο πολυσχηδεί, βλέποντας ότι η αλλαγή του κλίματος θα δημιουργήσει περισσότερες φυσικές καταστροφές στο μέλλον. Για να προστατεύσουμε καλύτερα τους πολίτες Χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, ούτω ώστε να προστατεύσουμε την Ευρώπη από τις φυσικές καταστροφές. Το RESC-EU είναι σχετικά καινούριο. Έχετε ήδη κάποια συμπεράσματα σχετικά με το πόσο αποτελεσματική είναι η εφαρμογή του ε, RESC-EU. Ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Το RESC-EU μόλις ξεκινάει Το χρησιμοποίησαμε το Rescue στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Εγώ θα εστιαζόμουν επί της εφαρμογής της διευρυσμένης συνεργασίας, του μηχανισμού διευρυμένης ε, πολιτικής προστασίας του Rescue. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τα αναγκαία μέσα στη διάθεσή της. Αυτό και η σαν πρόεδρος συμπεριέλαβε στο χαρτοφυλάκιό μου, στα καθήκοντά μου, στη σχετική επιστολή. Θα συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση αυτού. Θα συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσω ότι η διαδικασία προμηθειών θα ξεκινήσει ούτως ώστε να εξοπλιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μέσα που χρειάζονται. Αυτά τα μέσα είναι δαπανηρά, γι' αυτό υπάρχει σημαντικό ποσό που προβλέπετε, σημαντικό κονδύλι για πυροσβεστικά ε, αεροσκάφη, πυροσβεστικά ελικόπτερα, αλλά και δυνατότητες για ιατρική εκένωση και δυνατότητες για χημικά, πυρηνικά, βιολογικά προβλήματα και σχετικά μέσα ετοιμότητας για αυτά τα προβλήματα. Θέλω λοιπόν όλο αυτό το πακέτο να το υλοποιήσω, γι' αυτό θα εργαστώ. Αλλά πρωταρχικά το πρόβλημά μου θα είναι να πείσω τα κράτη-μέλη, αυτή θα είναι η πρόκληση, να τα πείσω τα κράτη-μέλη ότι αυτό είναι κάτι καλό, είναι προ όφελό τους, προ συμφέρον του και από την πρώτη μέρα αυτό προτίθεμαι να κάνω. Η συμπληρωματική ερώτηση. Ήδη αναφέρθηκε από κάποιο συνάδελφο και εσείς το θίξατε, αλλά θέλω να ρωτήσω αν έχετε συγκεκριμένες προτάσεις για περαιτέρω ενίσχυση της δυνατότητας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την πρόληψη φυσικών καταστροφών και των συνεπειών αυτών των φυσικών καταστροφών, η αντιμετώπιση άλλων απειλών, όπως είναι ατυχήματα που απαιτούν ιατρική υποστήριξη, χημικά ατυχήματα, πυρηνικά ατυχήματα, τέτοιου είδους ε, γεγονότα. Θα ήθελα να ρωτήσω επίσης κατά πόσο σχεδιάζετε να συνεργαστείτε με άλλους φορείς που υφίστανται για ταχεία αντίδραση. Δεν κατάλαβα το τελευταίο τμήμα της ερώτησής σας. Να συνεργαστώ με ποιον, ρωτήσατε. Μπορείτε να ξαναλάβετε το λόγο για να θέσετε το ερώτημα. Τελευταία φράση παρακαλώ, λέει ο υποψήφιος επιτροπός για το Κέντρο Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσης, ECBC. Αυτό πρέπει να το, το θεσμό πρέπει τον ερευνήσω. Δεν τον γνωρίζω αυτό το φορέα. Για τις δυνατότητες, για τον εξοπλισμό, πράγματι θα προσπαθήσω καταρχάς να εξασφαλίσω το ότι θα έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό ε, πυροσβεστικών αεροσκαφών. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Υπάρχουν κάποια και χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς το περασμένο καλοκαίρι στην Ελλάδα. Θα πρέπει να το συμπληρώσουμε αυτό και με πυροσβεστικά ελικόπτερα. Υπάρχουν και άλλοι δύο τομείς όπου το RESCUE eu πρέπει να είναι εξοπλισμένο με δυνατότητες για εκενώσεις ιατρικού ιατρικής φύσεως για θέματα χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά, πυρηνικά, για τέτοια ατυχήματα. Για τιμότητα και εξοπλισμό για τη μετώπιση αυτών των περιστατικών. Αυτά δεν είναι διαθέσιμα τα μέσα στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε αυτέ τι δυνατότητε, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αυτό το δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά αυτό εξαρτάται όμω από τα κράτη-μέλη, διότι τα κράτη-μέλη είναι εκείνα τα οποία αποφασίζουν περί τη ανάθεση και των διαγωνισμών για την απόκτηση αυτών των μέσων. Ο ρόλο μου είναι να πείσω τα κράτη-μέλη ότι αυτό είναι κάτι που είναι λογικό και έχει νόημα να το κάνουν. Ευχαριστώ. Λούκα Μάντελ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Λινάρτσος και καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ για την υποψηφιότητά σας ως νέο επίτροπο. Να μην ξεχνάμε ότι είναι πλεονέκτημα και προνόμιο να επιτελούμε σε τέτοια καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας έως τώρα. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ στην παρουσίασή σας είναι ότι αναφέρατε το σύμπλεγμα των εξωτερική δράση το οποίο θα ενταχθείτε στου κόλπους τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι όσο πιο πολλοί επίτροποι φροντίσουν για τι εξωτερικέ σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο καλύτερο. Και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ε, νομοθετούμε μόνο για το ιστορικό, θα πρέπει να ενισχύσουμε και το εξωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι τμήμα τη ε, αντίδραση στι εξωτερικέ κρίσει. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να σα ρωτήσω ποιο είναι ο συγκεκριμένο ρόλο σα αυτό το σύμπλεγμα θέσεων εξωτερικών υποθέσεων και πείτε μας για το σκέλος της πρόληψης όταν ε, κοιτάμε τη διαχείριση κρίσεων, φυσικών καταστροφέων, ενοπλών συγκρούσεων. Αν γίνει σωστή διαχείριση λοιπόν των κρίσεων στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φροντίσουμε δε και την σταθερότητα και την ειρήνη για να αποφύγουμε χειρότερες συγκρούσεις. Τι σκοπεύετε συγκεκριμένα να κάνετε για το σκέλος της πρόληψης. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων να έχει θέση και να συνεργάζεται με τους υπόλοιπους που ασχολούνται με την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνω, πρόκειται όμως για ένα τμήμα που από μόνο του στέκει και έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι ανεξαρτησία. Οι αποφάσεις όσον αφορά την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να λαμβάνονται ανεξάρτητα από τους άλλους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικούς, στρατιωτικούς, οικονομικούς, στρατηγικούς, οτιδήποτε. Αυτή η ανεξαρτησία είναι κάτι το οποίο θα υπερασπιστώ και όταν κάθομαι με τους υπόλοιπους της ομάδας για την εξωτερική δράση. Αλλά θα πρέπει να συντονιζόμαστε μεταξύ μας και προσβλέπω στην συνεργασία με τον το εκπρόσωπο τον κύριο Πορέλ με τον οποίο έχω ήδη συναντηθεί και ανταλλάξει απόψει και συμφωνώ μαζί σα για το ότι η πρόληψη είναι ακριβώ αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε. Γιατί είναι εύκολο να συνδυάσουμε ένα μεγάλο φάσμα μέσων εργαλείων που διαθέτουμε στην εξωτερική μας δράση με το στάδιο της πρόληψης. Και οικονομικά μας συμφέρει όπως καταλαβαίνετε. Κάθε ευρώ που επενδύουμε στην πρόληψη κρίσεων και καταστροφών μας εξοικονομεί κάπου 7 ευρώ που θα χρησιμοποιούσαμε αλλιώς για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης. Δεύτερη ερώτηση από τον ίδιο Ευρωβουλευτή. Ευχαριστώ. Πριν από δύο μέρες ε, εδώ πέρα είχαμε την κυρία Τουλάνεν που είναι η υπεύθυνη για διεθνή συνεργασία και είπε ότι ε, θέλει να συνεργαστεί μαζί σας ε, όσον αφορά την εκπαίδευση για τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, στους καταβλισμούς προσφύγων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ελπίζω θα ζητήσει πράγματι τη συνεργασία και ελπίζω αυτό να μην ε, πλήττει την ανεξαρτησία σας στην οποία αναφερθήκατε πριν. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια παρακαλώ για την ε, πολιτική προστασία. Γιατί είχαμε κατάσταση στην ε, προηγούμενη θητεία στις χώρες μέλη που ήταν πολύ διαφορετική από χώρα σε χώρα. Μπορείτε λοιπόν να το λάβετε υπόψη σας. Αυτό η κατάσταση είναι καλύτερη σε κάποιες χώρες και λιγότερο αλλού. Σίγουρα η ανεξαρτησία είναι πολύ σημαντική σε κάθε περίπτωση. Απάντηση. Ναι, ευχαριστώ. Σας διαβεβαιώ ότι θα συνεργαστώ με την συνάδελφό μου, την κυρία Ορπιλάινεν, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι ένας τομέας όπου οι εντολές μας, δεν θα λέγω ότι επικαλύπτονται, αλλά συναντιούνται. Ο δικός μου ο ρόλος είναι να διασφαλίσω ότι ακόμα και σε περιπτώσεις εκτεκτής ανάγκης, επίγουσες όπως τους καταβλισμούς προσφύγων, δεν παραβλέπουμε την εκπαίδευση. Μ' αρέσει αυτή η ιδέα. Εκπαίδευση σε επίγουσες καταστάσεις. Όπως είπα και πριν, όταν φτάνει ο Σεπτέμβριος, τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια πρέπει να γράφονται στα σχολεία. Ευχαριστούμε. Κύριε Κατρίν Σαμπόχη τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Μωριστέντε Επίτροπε, θέλω να επανέλθω λίγο στην σύνδεση της ανθρωπιστικής βοήθειας με την ανάπτυξη, αλλά να πάμε λίγο πιο μακριά στις φιλοδοξίες μας, κυρίως όσον αφορά τις νησιωτικές περιοχές που εκτίθενται όλος ιδιαίτερος εξαιτία τα μετρολογικά ακραία φαινόμενα πλήττουν αυτές τις περιοχές όλο και περισσότερο, όπως ήρμα και άλλα που έπληξαν διάφορες περιοχές. Στο σένα Μαρτά, η Ήρμα έκανε μεγάλες καταστροφές. Εγώ πήγα στο νησί, 1,5 χρόνο μετά τον ε, κυκλώνα, πήρε ε, βοήθεια το νησί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά, 1,5 χρόνο ακόμα τα σκουπίδια βρισκόντουσαν εκτεθειμένα και η ανοικοδόμηση δεν είχε προχωρήσει. Μιλώντας με τους διάφορους φορείς τοπικά, κατάλαβα ότι το δράμα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για να υπάρξει μια πραγματική αλλαγή στη σύνδεση της ανθρωπιστικής ε, βοήθειας με την βιώσιμη ανάπτυξη. Θα μπορούσε δηλαδή να βοηθήσει να γίνει και η ενεργειακή μετάβαση, η ενεργειακή αυτονομία, για αυτονομία όσον αφορά το νερό, ε, τα τρόφιμα κλπ. Οπότε η ερώτησή μου είναι εξή. Δεν Πιστεύετε ότι η διαχείριση κρίσεων θα μπορούσε να βοηθήσει ένα νησί για το μέλλον του και να αποτελέσει μια πραγματική στρατηγική για την βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών αλλά και για την αντίστασή τους και την αντοχή τους επόμενες κρίσεις. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου επιστήσατε την προσοχή στην κατάσταση αυτή σε ό,τι αφορά τα μικρά νησιά, τι νησιωτικέ περιοχές που αποτελούν περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες δεδομένε και της αλλαγή του κλίματο. Ξέρουμε ότι οι πάγοι στην Αρκτική και στην Αρκτική λιώνουν. Ξέρουμε ότι αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας και ξέρουμε ότι έχουμε διάφορα νησιά στην Καραϊβική και στον Νοτιοειρηνικό που θα αντιμετωπίσουν τεράστιες προκλήσεις. Αυτές οι χώρες έχουν περιορισμένους πόρους στη διάθεσή τους. Θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους και να τους βοηθήσουμε να προετοιμαστούν. Σε ό,τι αφορά γεγονότα και οι καταστάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να αποτρέψουμε, έχω για υπόψη μου για παράδειγμα τις ε, ε, ακραίε καιρικέ συνθήκε, την αύξηση τη στάθμης τη θάλασσα. Ξέρουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν και ότι θα χειροτερέψουν. Σημαντικό είναι να μην καθόμαστε με χέρια σταυρωμένα. Να βοηθήσουμε αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες, νησιωτικές χώρες, για να βελτιωθεί η κατάσταση ετοιμότητά του και η ανθεκτικότητά του. Εκεί θεωρώ ότι έχουμε ρόλο, όπω και έχει ρόλο και η συνάδελφο Ουρπιλάιεν με τον προπολογισμό για την ανάπτυξη. Για να βελτιωθεί λοιπόν η ανθεκτικότητα και η ετοιμότητα σε ό,τι αφορά την προσαρμογή στο κλίμα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τέτοια περιστατικά ή σε περιπτώσεις που γνωρίζουμε ότι είναι πιθανά διαφορά τέτοια περιστατικά. Ευχαριστώ πολύ. Ανα... Αναφερθήκατε στην αναγκαιότητα να στηριχθούμε στους τοπικούς παράγοντες σε ό,τι αφορά την βοήθεια αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι ε, παρούσα σε τέσσερις χρονιές του κόσμου. Σε ό,τι αφορά τη γεωστρατηγική λοιπόν αυτή η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να βρούμε τρόπους ε, ήδη για να βοηθήσουμε τις ΜΚΟ στις περιοχές αυτές για να υπάρχει καλύτερη ετοιμότητα σε ό,τι αφορά τα ακραία αυτά φαινόμενα προκειμένου να είναι πιο ταχεία για τη δρασή μας σε ό,τι αφορά τις καταστάσεις εκτάτου ανάγκη σε όλε τι άκρε του κόσμου. Χρειάζεται λοιπόν μια πραγματική στρατηγική για την βοήθεια σε αυτές τις περιοχές. Ο υποψήφιο επιτροπό Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Και συμφωνώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κινηθούμε. Να υπάρξει επιτόπου ανθεκτικότητα, να μην εστιαστούμε μόνο στην δυνατότητα ανταπόκρισης μας πρέπει να υπάρχουν και τα δύο σκέλη. Γιατί όταν χτυπήσει η καταστροφή χρειάζονται βοήθεια και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να την παρέχουμε. Δεν θα πρέπει λοιπόν να παραμελήσουμε καμία από τις δύο πλευρές. Ε, αλλά ναι, θα εργαστώ για την αύξηση της ανθεκτικότητας των ε, χωρών αυτών και μάλιστα θα συνεργαστώ στενά και με άλλους συναδέλφους, με άλλους επιτρόπους σε ό,τι αφορά το θέμα του περιβάλλοντος, των ωκεανών, της ανάπτυξης αναφέρθηκαν αυτά, γιατί όλοι θα πρέπει να συνεργαστούμε σε ό,τι αφορά αυτή την πράσινη συμφωνία τη Ευρώπη. Χρειάζεται πράσινη συμφωνία όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και για όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα μέτρα προσαρμογή στο κλίμα, τα μέτρα προετοιμασία, ετοιμότητα, προκειμένου είτε να αποφύγουμε, είτε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για τις καταστροφές αυτές. Ευχαριστώ. James Wells. Μη εγγεγραμμένος. Απουσιάζει. Νίκος Ανδρουλάκης για το S&D έχει το λόγο. Κύριε Πίτροπε, θέλω να σας ρωτήσω. Ε, εμείς μετά τις, φυσικές, μετά τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Σουηδία τα καλοκαίρια του 17 και του 18, ολοκληρώσαμε τον περασμένο Μάρτιο την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτική Προστασία. Δημιουργήσαμε λοιπόν έτσι το ΡΕΣΚΙΓΙΟΥ. Ακόμα όμω είμαστε σε μια μεταβατική φάση. Τα μέσα που βρίσκονται στη δεξαμενή ανήκουν αποκλειστικά στα κράτη-μέλη. Τώρα θα πρέπει να αποκτήσουμε τα ευρωπαϊκά μέσα. Αναφερθήκατε κι εσεί ότι η πρόκληση είναι η αντίδραση από τα κράτη-μέλη. Πώ θα διασφαλίσετε εσεί λοιπόν ότι το ΡΕΣΚΙΓΙΟΥ θα διαθέτει όλα τα αναγκαία μέσα για την καταπολέμηση των πυρκαγιών και άλλων καταστροφών και πώς σχεδιάζετε να ξεπεράσετε τα πιθανά εμπόδια ή την απορθυμία των κρατών μελών να αποκτήσουν αυτά τα αναγκαία μέσα. Επίση, ποια θεωρείται από αυτά ότι είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε ο μηχανισμό να είναι πλήρω λειτουργικό. Υποψήφια Επίτροπε. Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση που με επιτρέπει να αναλύσω περισσότερο το όλο θέμα. Ε, αυτό μου είπε η Πρόεδρος ότι ε, περιμένει να εξασφαλίσω, να εξασφαλίσω το ότι εντός του Rescue θα έχουμε ε, τα αναγκαία μέσα και σε επαρκή αριθμό τα μέσα αυτά. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν να διαθέσουν αυτά τα μέσα. Αυτό που έχω στη διάθεσή μου μόνο είναι τη δυνατότητα της πυθούς και ελπίζω ότι θα έχω και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να με βοηθήσετε πολύ σε αυτό το καθήκον, παροτρύνοντας τα κράτη-μέλη να διαθέσουν, να αγοράσουν αυτά, να αποκτήσουν αυτά τα μέσα. Δεν πρέπει να είναι τόσο δύσκολο. Πρέπει να πω ότι προσωπικά με κάπως βλέποντας αυτό τον αργό ρυθμό εφοδιασμού σε μέσα από τα κάτι μέλη. Γιατί, Γιατί εμένα μου φαίνεται πολύ καλή αυτή η συμφωνία. Από τη στιγμή που ένα κράτος μέλος Χ αποφασίζει να αποκτήσει ας πούμε πυροσβεστικά αεροπλάνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους κανόνες Rescue μπορεί να συγχρηματοδοτήσει μέχρι 90%. Οπότε βασικά σαν κράτος μέλος αποκτάς ε, για 10% της τιμής αυτό που θες μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το μόνο που υπογράφει είναι υποχρέωση όταν υπάρξει ανάγκη κάπου αλλού ότι θα πρέπει να διαθέσει αυτό το μέσο για να χρησιμοποιηθεί εκεί που υπάρχει η ανάγκη. Σαν απόθεμα ο το τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπαίνει στο αποθεματικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αυτό δεν ισχύει, το χρησιμοποιεί και το αποκτά στο 10% τη πραγματική τιμή. Η συμπληρωματική ερώτηση. Το 90% των χρημάτων για να αγοράσουν τα κράτη-μέλη τα εναέρια μέσα. Ε, θέλω επίση να σα ρωτήσω για το θέμα τη πρόληψη. Ε, είχαμε βάλει στο μηχανισμό την ανάγκη τα κράτη-μέλη να καταθέτουν και να μοιράζονται με την Επιτροπή τα σχέδια πολιτική προστασία, ώστε να τα αξιολογούμε και να βελτιώνονται. Εσείς θεωρείτε ότι αυτά τα οποία μέχρι σήμερα δίνουν ως στοιχεία για τους κινδύνους, για την προετοιμασία, για τον τρόπο αντιμετώπισης, είναι αυτά που χρειαζόμαστε ή πρέπει να μας δίνουν περισσότερα στοιχεία και συχνότερα και επίσης τι θα κάνουμε για να αναβαθμίσουμε αυτά τα σχέδια εθνική πολιτικής προστασίας ώστε να μειώσουμε τις φυσικές καταστροφές. Ε, ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση τα κράτη-μέλη όλα θα πρέπει κατά την άποψή μου να έχουν εφαρμόσιμα μέσα και στατηγικέ για τη μείωση των κινδύνων, διαχείριση των κινδύνων, στατηγικές γενικά και σύστημα, ε, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Και πρέπει να τα βοηθήσετε. Και εγώ είμαι έτοιμος ε, να βοηθήσω. Διότι η πρόληψη στον τομέα της πολιτικής προστασίας είναι η ευθύνη, εγώ προτιμώ τη λέξη ευθύνη, αντιαρμοδιότητα, responsibility and competence. Όταν μιλάμε για ευθύνη λοιπόν, δεν, δεν μπορεί να ο κόσμος αποκτήσει μεγαλύτερες ευθύνες, γι' αυτό μου αρέσει η λέξη ευθύνη, αντιαρμοδιότητα. Είναι ευθύνη λοιπόν των 100 η πολιτική προστασία και θα πρέπει αυτού του είδους αυτά να τα θεσπίσουν, να τα έχουν. Εγώ θα είμαι εκεί για να βοηθήσω, διότι έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε βέλτιστες πρακτικές από αλλού, έχουμε μηχανισμούς και εμπειρογνώμονες που μπορούν να βοηθήσουν και εγώ είμαι εκεί. Είμαι εκεί για να βοηθήσω τα κράτη-μέλη. Για να επομιστούν και να, εφαρμόσουν και να υλοποιήσουν αυτές τις ευθύνες. Δίνω το λόγο στην Λουτμίλα Νοβάκα από το ΕΛΚ. Κύριε υποψήφιε Επίτροπε Γιάννη Λένατσικ, σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω να μου απαντήσετε στα σλοβενικά, στη μητρική σας γλώσσα συζητήσαμε το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευαίσθητη σε ό,τι αφορά τι ανάγκε των ανθρώπων που τη χρειάζονται και στι χώρε που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκη και είναι μία από τι μεγαλύτερε δωρήτριε. Και σκοπό μα είναι να αυξήσουμε αυτή την βοήθεια. Πιστεύετε ότι το σύστημα διανομή τη βοήθεια μέσω των ΜΚΟ είναι αρκετά διαφανέ, αρκετά αποτελεσματικό και έχει μακροπρόθεσμα θετικέ επιπτώσει. Δυστυχώ, ακούμε συχνά από διάφορες, ε, ότι διάφορες μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις σε ό,τι αφορά την αναδιανομή των πόρων τελικά χρηματοδοτούν οργανώσεις οι οποίες δεν λειτουργούν βάσει των ευρωπαϊκών ε, αρχών. Θα αναβαθμίσετε το σύστημα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Η απάντηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε να απαντήσω στη μητρική μου γλώσσα. Ασφαλώς και είναι δικαίωμά μας. Χάρη στην υπηρεσία διερμηνίας. Εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειριζόμαστε την ανθρωπιστική βοήθεια βάσει της συνεργασίας με τις ε, οργανώσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε, η υποτερμοστία του ΟΗΕ και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις αφετέρου. Πιστέψτε μας, κάνουμε εντελεχή έλεγχο για να καθορίσουμε κατά πόσον οι οργανώσεις αυτές μπορούν να λειτουργήσουν και λειτουργούν όπως πρέπει. Και θα πρέπει να τηρούν ε, ε, διάφορες αρχές, ε, η αμεροληψία, η διαφάνεια, ανθρωπισμός. Και μία άλλη αρχή η οποία είναι δύσκολο να την ε, μεταφράσω από τα αγγλικά τα οποία συνήθως ε, χρησιμοποιώ θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι αυτά τα χρήματα οικονομικά μέσα τα οποία διατίθενται είναι χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Για ποιον λοιπόν προορίζονται αυτά τα μέσα, για ποιο σκοπό, για να σωθούν οι ζωέ των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ελέγχουμε και ελέγχουμε πάρα πολύ προσεκτικά κατά πόσον οι εταίροι μα πραγματικά διαχειρίζονται σωστά τα μέσα αυτά για να μην σπαταλώνται αυτά τα χρήματα, αυτή η πόρη. Και για να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα αυτά χορηγούνται προς το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Και για να υπάρχει πραγματικά καλή παρακολούθηση των κονδυλίων αυτών, να δούμε πώς ε, δαπανώνται. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Συμπληρωματική ερώτηση. Δεν χωράει αμφιβολία ότι γνωρίζετε μάλλον ε, την Πέτρα Πέκ, η οποία είναι ιεραπόστολο στην ε, Μαλασκάρη. Έχει διδάξει τους ανθρώπους εκεί πώς ε, να ψαρεύουν και έτσι δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο χωριό σε μια περιοχή λιμάτων. Κατάφερε λοιπόν να βοηθήσει και να διδύσει ένα ολόκληρο σύστημα, ένα ολόκληρο χωριό και έτσι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια δουλειά και μπορούν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό του. Και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώ μπορούμε να παρέχουμε βοήθεια σε κόσμους, στον κόσμο σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Μιλήσατε για τι τοπικέ ε, ανάγκες, τις ανάγκες επιτόπου. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό μπορούμε να δείξουμε στον κόσμο επιτόπου πώς μπορεί να λάβει υποστήριξη και μάλιστα με προληπτική με προληπτικό τρόπο, προκειμένου να αναπτύξουν διάφορε τέτοιε δραστηριότητε. Ο υποψήφιο επιτροπό. Το έργο. Του Ιεραπόστολου αυτό το γνωρίζω πολύ καλά και στο τοπικό επίπεδο μπορούν πολλά να γίνουν για να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια στην ε, ρίζα τη. Και τα υποστηρίζουμε αυτά προφανώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν ε, επιβεβαιωθώ στη θέση μου ως Επιτροπός, δεν θα είμαι άμεσα αρμόδιος για τέτοια ζητήματα, αλλά σε ό,τι αφορά το προληπτικό σκέλος των δράσεών μας, και σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της ανθεκτικότητας ε, της ε, κοινότητας ε, αυτής που αναφέρατε, σε ό,τι αφορά και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, γιατί πολλοί από τους στόχους αυτούς μπορούμε να τους πετύχουμε μόνο αν αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τις ανθρωπιστικές κρίσεις ή αν υπάρχει πρόληψη των κρίσεων αυτών Το έργο του Ιεραπόστολου ΟΠΕΚΑ αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην πρόληψη, στο σκέλος της πρόληψης ανθρωπιστικών κρίσεων και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιτήτων και κοινωνιών. Και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων και σέβομαι το έργο του. Like the... Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μανών Ομπρή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να αναφερθώ και εγώ σε κάτι το οποίο ήδη συζητήσαμε κάπως, αλλά ήδη αυτή τη βδομάδα σήμερα ο πρόεδρος της Action Securité κλήθηκε από τις αρχές εσωτερικής ασφάλειας στη Γαλλία επειδή κατάγγειλε την εξαγωγή όπλων από τη Γαλλία στην Ιεμένη. Λοιπόν, δεν είναι κανένα μυστικό αυτό, αλλά είναι μια υποκρισία αυτή Συνεπώς, στέλνουμε ανθρωπιστική βοήθεια ε, σε κάποιες χώρες, στις οποίες εξάγουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπλα, με αποτέλεσμα βέβαια να χάνονται πολλές ζωές. Η Εμένη, όπως το είπατε και εσείς, βρίσκεται σε μία από τις χειρότερες κρίσεις που έχουμε σήμερα στον κόσμο. Οπότε, Έχουμε εξαγωγή όπλων, τεχνολογίας πολεμικής από πλευρά στο χωρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα λάβουμε υπόψη μας λοιπόν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς θα συντονίσετε την Ευρωπαϊκή Ανθρωπιστική Βοήθεια με την αυστηρή εφαρμογή των ε, όσων ισχύουν για αυτήν. Απάντηση. Αναφέρατε αξιότιμη Ευρωβουλευτή, την ε, εξογωγή όπλων. Κοίταξε, όσον αφορά την αρχή, συμφωνώ. Οι ανθρωπιστικές κρίσεις συχνά, όχι πάντα, εν μέρη τουλάχιστον, δεν ε, είναι συνέπεια μόνο μιας εμπόλεμης ε, σύγκρουσης, όπου χρησιμοποιούνται φυσικά όπλα και πράγματι πολλές χώρες κάνουν εξαγωγή όπλων. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα μέσα στην οποία πρέπει να δράσουμε κι εμείς. Φυσικά και πρέπει να δώσουμε σημασία σε αυτό το θέμα της εξαγωγής σε περιοχές του κόσμου που υπάρχουν συγκρούσεις. Υπάρχουν προδιαγραφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να τηρούνται για παράδειγμα στην εξαγωγή όπλων, να μην δρούμε με τρόπο που θα επιδίνωνε την ανθρωπιστική κατάσταση. Και νομίζω ότι είναι το καθήκον, θα είναι το καθήκον μου εφόσον επιβεβαιωθώ ε, στην ε, θέση αυτή, να τονίσω και να υπογραμμίσω ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς στη συμπεριφορά μας. Δεν πρέπει να εξάγουμε δηλαδή όπλα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιδεινώνονται ανθρωπιστικές κρίσεις. Ε, δεύτερη ερώτηση. Ακούω τη δέσμευσή σας. Ναι, και ευχαριστώ. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τον το ρόλο που παίζουν οι χώρες μέλη όταν εξάγουν σε τέτοιες χώρες και τις επιπτώσεις στην ανθρωπιστική κρίση εκεί. Ακούω λοιπόν την προφορική σας δέσμευση. Πέρα από αυτό, σκοπεύετε να στείλετε ένα ισχυρό μήνυμα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάτε και πιο μακριά και να κάνετε πραγματικότητα αυτό που ζητάνε πολλέ διεθνεί οργανώσει, μεταξύ άλλων και Amnesty International, για εμπάργκο όπλων προς χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη σύγκρουση. Γιατί έτσι παραβιάζεται το ανθρωπιστικό δίκαιο και επιδεινώνεται η κατάσταση σε χώρες όπως για παράδειγμα η Εμένη. Ο Επιτροπός, υποψήφιος Επιτροπός. Σκοπεύω να συνεργαστώ με τους υπόλοιπους Επιτρόπους προκειμένου να το κοιτάξουμε αυτό το θέμα περισσότερο σε βάθος. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ναι. Πρέπει να υπάρχει μία αρχή που να τηρούμε. Δηλαδή, όταν υπάρχει εμπόλεμη σύγκρουση, εμείς να προσέχουμε πολύ καλά τι κάνουμε και όσον αφορά την εξαγωγή όπλων. Μπορεί να αποφεληθεί από αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σωστά είναι περήφανη για το γεγονός ότι είναι ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά αν από την άλλη μεριά κάνουμε πράγματα τα οποία επιδεινώνουν την ανθρωπιστική κρίση, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν αρμοδιότητες και ευθύνε και κάποιες από αυτές βρίσκονται στα χέρια των χωρών πελών. Αλλά σας μίλησα για την αρχή που πρεσβεύω. Και αυτό που είπα εδώ θα το πω ξανά, ότι οι δράσεις μας δηλαδή πρέπει να είναι συνεπείς. Πρέπει να αποφεύγουμε την επιδίνωση ανθρωπιστικών κρίσεων μέσω των ε, δράσεών μας ε, στον τομέα της εξαγωγής όπλων. Αλλά δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση που εξάγει τα όπλα, έτσι. Είναι οι χώρες μέλη. Ναι. Ευχαριστώ. Ιζαμπέλ Σάντος για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, έχουμε πολλές συγκρούσεις στον κόσμο, έχουμε το, την κρίση του κλίματος, όλο και περισσότερες προκλήσεις όσον αφορά το επίπεδο και την ποιότητα της ανταπόκρισής μας και το τι κάνουμε εξασφαλίσουμε ότι γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ανταποκρισή μας. Άκουσα πολύ προσεκτικά και σημείωσα την πρόθεσή σας να συμμετέχουν περισσότερο οι ΜΚΟ συμπεριλαμβανομένων των τοπικών φορέων των ΜΚΟ. Και αυτό ευθυγραμμίζεται ε, με τη δουλειά που κάνατε σαν επικεφαλής στον ΤΥΡ. Σας παρακολουθούσα τότε που προασπίζατε τους ακτιβιστές και αυτά που έκαναν επί τόπου. Λοιπόν, και εκεί υπήρχε αυξανόμενη συμμετοχή των ΜΚΙΟ. Χρειάζεται πάντα αποτελεσματική ανταπόκριση υψηλή ποιότητα. Μιλήσατε για τη μεγάλη συμφωνία, το Grand Bargain. Τι γίνεται με τη διαφάνεια όμω σε αυτό το τομέα. Και για το συντονισμό Θέλω να μου πείτε περισσότερα για συντονισμό. Όταν έχουμε κατεπίγουσα ανάγκη επιτόπια και ανταποκρινόμεθα ανθρωπιστικά, συχνά βλέπει κανείς ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού. Και σπαταλώνται πολλοί πόροι. Πώς θα βελτιώσετε λοιπόν την ποιότητα του συντονισμού που απαιτείται. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, η απάντησή σας. Ευχαριστώ κυρία Σάντος. Μεγάλη χαρά για μένα να σας βλέπω εδώ. από την παλιά μας θέση βρεθήκαμε τώρα στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλη χαρά που σας βλέπω εδώ ξανά. Ο συντονισμός είναι πάντα πρόκληση. Όταν έχει πάρα πολλούς φορείς, όπως σε διεθνή ανθρωπιστική ε, βοήθεια, υπάρχουν πολυπληθείς οργανώσεις, φορείς, ΜΚΟ, Υπάρχουν κάποιες προφανείς λύσεις. Υπάρχουν και κάποιες αρχές που ακολουθούμε και λειτουργούν καλά κανονικά. Να συμφωνήσουμε καταρχάς ότι ο ΟΗΕ και πιο συγκεκριμένα το γραφείο του ΟΗΕ για συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων θα πρέπει να έχει το ρόλο του γενικού συντονισμού. Το υποστήριζα και το υποστηρίζω αυτό. Θα είναι ένα από τα πρώτα μου βήματα αν εγκριθεί ο διορισμός μου. Να έρθω σε επαφή με τον ΟΗΕ και την υπηρεσία αυτού για συντονισμό των ανθρωπιστικών υποθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως επίσης πρέπει να ασταλάξει το πνεύμα συντονισμού και συνεργασίας. Να ξέρουν όλοι τι θα κάνει, όλοι να γνωρίζουν τα καθήκοντά τους σε μια ανθρωπιστική επιχείρηση. Θα ήταν σπατάλη ατυχής αν στον τομέα όπου έχουμε τέτοια χρηματοδοτικά κενά να σπαταλήσουμε πόρους λόγω ελλείψεως συντονισμού. Συμβαίνει, το γνωρίζω αυτό, υπήρξαν περιπτώσεις κατά το παρελθόν, όπως πριν πολλά χρόνια στην ΑΕΤ και αλλού, αλλά θα πρέπει να παλέψουμε ούτως ώστε να σταλάξουμε κάποια πειθαρχία και να αναγνωρίσουμε το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών που θα πρέπει να έχει το γενικό συντονισμό, να έχουν το γενικό συντονισμό και να μοιραστούμε μεταξύ μας τα καθήκοντα. Με έναν τρόπο που θα είναι συνεργατικός και συντονισμένος. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναφερθήκατε Ανθεφερθήκαμε εδώ στην ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί στους προσφυγικούς καταβλισμούς στη Λέσβο. Προσπαθήσαμε να μειώσουμε τη ροή των μεταναστών και συνάψαμε συμφωνία με τη Λιβύη. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση στη Λιβύη. Όλοι γνωρίζουμε όσον αφορά του μετανάστε και του πρόσφυγες και όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά την κατάσταση που επικρατεί στα κέντρα α, ε, των προσφύγων στη Λιβύη. Από πλευρά ανθρωπιστική είναι απέσια, φρικτή κατάσταση που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα κάποιο σχόλιο σα πάνω σε αυτό. Και πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, απάντηση. Σα ευχαριστώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η κατάσταση στα κέντρα κράτηση ε, είναι φρικτά στη Λιβύη. Φρικτά, απέσια κατάσταση. Προσπαθεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε εκεί. Έχουμε ανθρωπιστικά προγράμματα για παροχή βοήθειας η κατάσταση όμως αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μετακινηθούν, να φύγουν από αυτά τα κέντρα και να πάνε αλλού. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να μετεγκατασταθούν. ή κυρίως εκείνοι που δεν έχουν δικαίωμα διεθνούς προστασίας να βοηθηθούν να επιστρέψουν στην χώρα καταγωγής τους. Αλλά συμφωνώ, πράγματι. Είναι πολύ κακή η κατάσταση. Και η ανθρωπιστική βοήθεια δεν αποτελεί λύση. Όπως είπα ήδη, η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι εργαλείο διαχειρίσεως των κρίσεων. Δεν λύνει τις κρίσεις. Προσπαθεί να καλύψει τις άμεσες ανάγκες των πληγέντων πληθυσμών. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στα κέντρα κράτησης στη Λιβύη. Περισσότερα πρέπει να γίνουν. Συμφωνώ. Να βρούμε πιο βιώσιμες λύσεις γι' αυτό. Σας ευχαριστώ και τώρα να δώσω το λόγο στην ε, Αλεξάνδρα Λουίς Ρόζενφελ ε, από τους Πράσινους. Ξέρω ότι σας έχουν θέσει παρόμοιες ερωτήσεις ε, και ως Επίτροπος Αντιμετώπισης των Κρίσεων θα εργαστείτε για το κόστος της απραξίας. Ξέρετε πως οι άνθρωποι θα μπορούσαν να χρειάζονται ε, ανθρωπιστική βοήθεια μέχρι το 2030 λόγω φυσικών καταστραφών, μέχρι το 2050, αν δεν δράσουμε τώρα σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την ε, αλλαγή του κλίματο. Αν δεν λάβουμε λοιπόν μέτρα τώρα, ο αριθμό των ανθρώπων που θα χρειάζεται κάθε χρόνο ε, ανθρωπιστική βοήθεια μέχρι το 2050 θα διπλασιαστεί κάθε χρόνο και θα φτάσουμε τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε ανθρωπιστική βοήθεια που θα χρειάζεται. Αυτό το σενάριο όμως μπορούμε να το αποφύγουμε αν επενδύσουμε σε προσαρμογή στο κλίμα και μείωση στις αλλαγές του κλίματος, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων που είναι σε κίνδυνο και βελτιώνοντας ε, τις δράσει για την έγκυρη προειδοποίηση. Πώς θα ενσωματώσατε λοιπόν μια πιο πράσινη προσέγγιση στον τομέα τη ανθρωπιστική βοήθεια και τι συγκεκριμένα μέτρα θα πάρετε προς το σκοπό αυτό. Τι κονδύλια θα κινητοποιήσετε για να ανταποκριθείτε σε τέτοιε φυσικέ καταστροφέ. Ευχαριστώ. Ο υποψήφιο επιτρόπο για να απαντήσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντική ερώτηση αυτή και θα στραφώ στο σημείο που ξεκίνησα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εναρμονίσουμε την μείωση του κινδύνου από καταστροφές και όλο αυτό να μπει μέσα στην Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη και τη συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το κόστος της απραξίας θα είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με αυτά που πρέπει να κάνουμε για να αποτρέψουμε ή να μειώσουμε τον αντίκτυπο περιστατικών που δεν μπορούμε να αποτρέψουμε πλήρως. Και θα εργαστώ επ' αυτού. Θα συνομιλήσω και με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο, τον κύριο Τίμερμαντς, για να συμπεριληφθεί ο κίνδυνος και η στρατηγική για τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών σε όλες τις δράσεις για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό η κατάσταση με την οποία θα είμαστε αντιμέτωποι θα είναι πολύ χειρότερη και θα είμαστε απροετοίμαστοι. Και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επενδύσουμε πολύ παραπάνω από αυτά που καλούμαστε να επενδύσουμε τώρα. Ένα ευρώ στην πρόληψη μας ε, εξοικονομεί μέχρι και 7 ευρώ στην αντιμετώπιση μιας κατάστασης που θα μπορούσε να έχει προβληθεί. Η συμπληρωματική ερώτηση. Μάλιστα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας. Είπαμε σήμερα το απόγευμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να αυξήσει τη συμμετοχή του δυτικού κλάδου σε ό,τι αφορά τις δράσεις της. Ωστόσο, υπάρχουν όροι προκειμένου να παραμείνουν στα ίδια πρότυπα και ιδιωτικό κλάδο όπω και η διεθνή ΜΚΟ ο ιδιωτικό κλάδο λοιπόν που θα συμμετέχει σε τέτοια έργα ανθρωπιστική βοήθεια, πώ θα εξασφαλίσετε ότι θα τηρήσει τα ίδια πρότυπα σε ό,τι αφορά το διοξείδιο του άνθρακα, τι εκπομπέ αερίου του θερμοκηπίου. Οι εταιρείε οι οποίε ρηπαίνουν και οι οποίε είναι υπεύθυνε σε μεγάλο βαθμό για την μόλυνση τη ατμόσφαιρα ε, θα πρέπει να συμβάλλουν σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Ευχαριστώ πολύ. Η απάντηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να συνεργαστούμε με τον δυτικό κλάδο και ιδιαίτερα ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος και το σώμα των επιτρόπων δεν θα είναι σε θέση να πετύχει όλες τις πτυχές του, της Πράσινης Συμφωνίας για την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο αν δεν συμμετέχει και ο δυτικό κλάδος για τον πολύ απλό λόγο ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις που χρειάζονται για να μπορέσει αυτή η πράσινη συμφωνία, το Green Deal, να πραγματοποιηθεί και αυτό ισχύει και για τα μέτρα προετοιμασίας και πρόληψης που θεωρώ ότι εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιό μου γιατί έχουν να κάνουν με τον κύκλο διαχείρισης κρίσεων Διαχείριση κρίσεων. Περιμένουμε να χτυπήσει το τηλέφωνο, να το σηκώσουμε και να απαντήσουμε, να διαχειριστούμε μια κρίση. Η ετοιμότητα και η προετοιμασία και η πρόληψη είναι πιο σημαντικά σκέλη. Πιο σημαντικά γιατί είναι και πιο φθηνά. Μιας και έχουμε λοιπόν περιορισμένους πόρους, θα καλύτερα θα τα κάναμε να επενδύσουμε σε αυτόν το σκέλος. Θα συνεργαστώ λοιπόν με τους επιτρόπους ε, συναδέλφους μου που είναι αρμόδιοι για θέματα κλίματος, ε, περιβάλλοντος, ωκεανούς κτλ. Γιατί η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί κοινή ευθύνη, κοινό στόχο και σκοπεύω να συμβάλλω με τον τρόπο που περιγράψατε. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Βερονίκ Τριγέλη Νουάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Οριστέντα Επίτροπο. Σήμερα πάνω από 80% του κόσμου απειλείται από διάφορες ε, μεταδοτικές ασθένειες. Και τώρα αυτό έχει να κάνει και με την Ευρώπη. Και ίσως οφείλεται το φαινόμενο αυτό, λένε πολλοί, στις μεταναστευτικές ροές, κάτι το οποίο όμως επιστημονικά δεν στέκει. Και άλλοι λένε ότι το θέμα αυτό έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή και την θέρμανση του πλανήτη και όχι με τις μεταναστευτικές ροές. Τώρα λοιπόν, επιδημίες, ελονοσία, τσιτσιγκούνια, πυρετός, τέγκια κτλ. εμφανίζονται στην Κροατία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στη δικιά μου τη χώρα, τη Γαλλία. Οπότε κύριε Ριστέντα, Επίτροπε, αυτό μπορεί να αποτελέσει σημαντική απειλή στο μέλλον. Πώς θα προστατεύσετε εσείς τους Ευρωπαίους λοιπόν από αυτές τις νεοαφιχθήσεις ασθένειες. Ο οριστής Επίτροπος, ευχαριστώ για την ερώτησή σας αυτή. Νομίζω ότι η απειλή είναι πραγματική και έχει βάση αυτό που λέτε. Η απειλή δηλαδή τέτοιων μεταδοτικών ε, ασθενειών που μεταφέρονται δηλαδή από φορείς είναι μια πραγματικότητα. Και δεν είμαστε έτοιμοι, καθόλου δεν είμαστε έτοιμοι. Και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε. Γιατί ασθένειες που κάποτε ήταν χαρακτηριστικό τροπικών χωρών και περιοχών του κόσμου, και μόνο όταν ταξιδεύαμε σε εξωτικά μέρη κινδυνεύαμε από αυτές, τώρα έρχονται στις χώρες μας. Και δεν έρχονται στις χώρες μας από ανθρώπους, αλλά από έντομα. Αν λοιπόν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, εγώ θα συνεργαστώ με την Στέλλα που είναι υποψήφια επίτροπος υγείας και θα κοιτάξουμε πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα. Εκείνη θα έχει στη διάθεσή της όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής που μπορούν να βοηθήσουν στον τομέα της υγείας και εγώ από τη δικιά μου την πλευρά μπορώ να συνεσφέρω με τον συντονισμό της ε, βοήθειας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προετοιμαστούμε. Και πρώτα απ' όλα μπορούμε να αναπτύξουμε εμβόλια. Ε, μπορούμε επίσης να τα αποθηκεύσουμε για την περίπτωση που θα έχουμε κάποια επιδημία. Αν ξεσπάσει δηλαδή μια επιδημία. Και μία επιλογή θα ήταν ο μηχανισμός Rescue θα μπορούσε δηλαδή να αποθηκεύει τέτοια εμβόλια για την περίπτωση που έχουμε ξέσπασμα μιας τέτοιας ασθένειας. Συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ τον ε, οριστέντα επίτροπο για την τόσο ειλικρινή και τίμια απάντησή του ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι και ακριβώς και εγώ αυτό θα ήθελα να προειδοποιήσω ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι προτείνω να δουλέψετε επίσης και πάνω σε συστήματα προειδοποίησης. Να προειδοποιούνται και όσοι εργάζονται στην υγεία, αλλά και γενικότερα ο κόσμος για την έλευση τέτοιων ασθενειών. Ευχαριστώ. Ο οριστής επίτροπος. Ναι. Ναι, θα το κάνω. Σε στενή συνεργασία με την Επίτροπο την Αρμόδια για θέματα υγείας. Σας ευχαριστώ για τελευταία ερώτηση. Francis Fitzgerald από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Καλή αργά παρά ποτέ. Καλησπέρα υποψήφια Επίτροπε. Άλλη μια ερώτηση για ένα βασικό θέμα που έθεσαν πολλοί συναδελφοί μου. Από ό,τι καταλαβαίνω, από την ανάθεση του χαρτοφυλακίου σας. Ο ρόλος σας στη διαχείριση των κρίσεων είναι ένας ρόλος πρόληψης και μείωσης των συνέπειων. Και είναι σαφές που, όπως είπαν συναδέλφοι, τα τελευταία χρόνια πραγματικά γεγονότα όπως οι καταστροφικοί κυκλώνες, οι δασικές πυρκαγιές κλπ. Βλέπουμε ότι η αλλαγή του κλίματος έχει δημιουργήσει αυτές τις καταστροφές και έχουμε αυτές τις συνέπειες. Ερώτηση. Πώς θα ενσωματώσετε προληπτικά και μέτρα και μέτρα μείωση των συνεπειών όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και αντοχή στην αλλαγή του κλίματος. Στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης, σε συνεργασία με τους συναδέλφους σας επιτρόπους, διότι πιστεύω ότι όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να συνεργάζονται οι επίτροποι. Πέρα από τα όρια των χαρτοφυλακίων τους να κινούνται ε, ενωμένοι. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε. Ευχαριστώ το αξιότιμο μέλος για αυτή την ερώτηση. Πράγματι, περί αυτού πρόκειται. Δεν νομίζω ότι οσδήποτε επίτροπος μόνος του ή μόνη της είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Θα είναι ιδιαίτερο πρόβλημα και πρόκληση για το μελλοντικό σώμα των επιτρόπων να βρουν έναν τρόπο αποτελεσματική συνεργασία από αυτόν. Από την πλευρά μου βλέπω μια ιδιαίτερη δυνατότητα να τροφοδοτώ εγώ τους την εργασία των άλλων μέσω πρόληψης και όταν δεν υπάρχει άλλη λύση προσαρμογή. Πώς λειτουργούν αυτά. Ας προσπαθήσω να εξηγήσω. Ήδη σήμερα μιλήσαμε για το Σαχέλ και το κέρας της Αφρικής. Είναι περιοχές που ήδη αισθάνονται τον αντίκτυπο της αλλαγής του κλιμάτος. Οι βροχοπτώσεις άλλαξαν αυξήθηκαν οι περίοδοι της ξηρασίας, οι περιοχές που υφίστανται αυτή την ξηρασία. Τι κάνουμε λοιπόν για να προσαρμοστούμε. Ένας τρόπος είναι να δούμε τις οδιές που παραδοσιακά καλλιεργούνται και να δούμε κατά πόσο μπορεί να αντικατασταθούν με κάποιες άλλες οδιές, άλλα προϊόντα που να αντέχουν περισσότερο στην ξηρασία και τη ζέστη δεν είναι κάτι που αποφασίζω εγώ σαν μελλοντικό επίτροπος, αλλά οι συνάδελφοι ανάπτυξη θα αποφασίσουν σε συνεργασία με τους ειδικού για τη γεωργία που γνωρίζουν την περιοχή. Ούτω ώστε να έχουμε αποτελεσματική πρόληψη και προσαρμογή πρέπει να συνεργαστούμε. Πρώτα απ' όλα εντό τη Ευρωπαϊκή επιτροπή αλλά μετά και με του εταίρου μα εντό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω Έτσι θα είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά μέτρα για να αποφύγουμε και να μειώσουμε, όπως είπατε, να μειώσουμε τον αντίκτυπο ε, της αλλαγής του κλίματος. Συμπληρωματική ερώτηση. Αναφέρθηκα σε συνεργασία πέρα από τα χαρτοφυλάκια τα ξεχωρισμένα, αλλά ήδη αναφερθήκατε, καλύψατε κάπως και τη δεύτερη ερώτησή μου, δηλαδή να τονίσουμε την ανάγκη συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών, με ΜΚΟ και να δημιουργηθούν ισχυρές συνεργασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά και στις σχέσεις με τρίτες χώρες, στο επίκεντρο των προσπαθειών και διαδικασιών να μπουν οι πολίτες. Θα χρειαστούμε αυτά τα στοιχεία που προανέφερα ακόμα πιο ανεπτυγμένα από ό,τι είναι στο παρόν, επί του παρόντος. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, ναι, συμφωνώ. Σωστό αυτό. Πρέπει να συμμετάσχουν και οι ΜΚΟ. Όλες αυτές οι προσπάθειες θεωρώ ότι είναι σημαντικό τμήμα της φιλοδοξίας μας να πετύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Η στρατηγική για επίτευξη των στόχων είναι αυτή. Να συμμετέχουν όλοι οι φορείς και η ΜΚΟ είναι σημαντική φορή κυρίως στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Έχουμε πολύ θετική εμπειρία από τη συνεργασία μας με τις ΜΚΟ. Είναι εταίροι μας αξιόπιστοι που τι εμπιστευόμεθα, αποτελεσματικοί εταίροι. Είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς αυτή η συνεργασία μπορεί, τι μορφή μπορεί να έχει και θα έχει, ούτω ώστε από κοινού να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τις ερωτήσεις που έκαναν και ασφαλώς και τον υποψήφιο επίτροπο για τις απαντήσεις του. Okay, we just have a question now going to allow another το θέμα του κατά πόσον θα επιτραπεί μια επιπλέον ερώτηση. Θα σας δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρα και σας ευχαριστώ υποψήφια Επιτροπέ. Δεν θέλω να σας ε, κάνω να αισθανθείτε αδικημένος, γιατί είχαμε μόνο 24 ερωτήσεις, γιατί ένα μέλος δεν ήρθε στην ακρόαση με την ε, έγκριση και την άδεια του Πρόεδρου. Θα ήθελα να θέσω άλλη μία ερώτηση. Ο Πρόεδρος, έχουμε ήδη διαιρέσει το χρόνο μεταξύ των πολιτικών ομάδων και σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένου, οπότε... Δεν θα επιτρέψω την ερώτηση και ζητώ συγγνώμη. Δεν θέλω να γίνω κακό, αλλά σε κάποιε περιπτώσει πρέπει να τηρούνται οι κανόνε και ξέρω ότι έχουμε πολλέ ερωτήσει από την Επιτροπή, τι συνδεδεμένε επιτροπέ και γι' αυτό θα δείξω μια έμονη στου κανόνε στο σημείο αυτό και θα ήθελα να ανακοινώσω το εξή. Θα συναντηθώ με του ε, συντονιστές για να κάνουμε αξιολόγηση της ακρόασης και κλεισμένων των θυρών, όπως ξέρετε. Ξέρετε πότε θα λάβει η χώρα αυτή η συνεδρίαση. Να πω ξεκάθαρα ότι δεν θα μπορέσετε να στείλετε οποιονδήποτε ε, πολιτικό σύμβουλο για να σας αντικαταστήσει. Μόνο τα μέλη της Επιτροπής μπορείτε να πάρετε μαζί τους βοηθούς σας, αλλά δεν θα μπορούν να σας αντικαταστήσουν στη συνεδρίαση αυτή. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο, στον υποψήφιο Επίτροπο μάλλον, για να κάνει τα καταληκτικά του σχόλια. Έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ τους αξιότιμους ευρωβουλευτές για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε, για την ευκαιρία δηλαδή που μου δώσατε. Πραγματικά ήταν κάτι που με κράτησε σε γρήγορη συνέχεια. Χάρηκα τη συζήτηση αυτή μαζί σας. νομίζω ότι σε ένα βαθμό μπόρεσα να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Επιτρέψτε μου να πω επίσης ότι στην περίπτωση που επιβεβαιωθώ για την θέση του Επιτρόπου, νιώθω ήδη το βάρος της ευθύνη του ώμους μου. Δεν παίρνω καθόλου στα ελαφρά το χαρτοφυλάκιό μου. Είναι μια ευγενής αποστολή είναι ένας τρόπος για να δείξουμε την καλύτερη εικόνα της Ευρώπης και εκτός Ευρώπης και μέσα στην Ευρώπη. Η αλληλεγγύη είναι κάτι που δεν σκέφτεται ο κόσμος μέχρι τη στιγμή που θα τη χρειαστεί και τότε τη θυμούνται για πάντα. Θα ήθελα λοιπόν, εφόσον επιβεβαιωθώ σε αυτή τη θέση, να συνεργαστώ στενά μαζί σας για να χτίσουμε μαζί μια συνεργασία, εταιρική σχέση που υπάρχει παραδοσιακά βέβαια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μια τελευταία παρατήρηση για την επιστολή ανάληψης καθηκόντων για το χαρτοφυλάκιό μου. Κάποιος κάτι με ρώτησε για το πρώτο θέμα που έβαλε στην επιστολή αυτή η νέα πρόεδρος και ήταν αυτό το κέντρο συντονισμού το οποίο εγώ θα το ενισχύσω ακόμα περισσότερο Πάντως, μπορεί να μην απάντησα πριν, αλλά τώρα θα σας πω ότι είναι κάτι υπέροχο. Εγώ το επισκέφτηκα και αν δεν το έχετε επισκεφθεί ακόμα, είναι εντυπωσιακό και είναι και εντυπωσιακό προς τον έξω κόσμο. Γιατί αυτό το κέντρο ανταποκρίνεται στις αιτήσει που έρχονται για βοήθεια, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Οπότε ε, θα ρωτήσω και εγώ αυτό που ρώτησε ο Χένρι Κίσιγκερ κάποτε. Ποιο είναι το τηλέφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, λοιπόν, αν πρόκειται για επίγουσα βοήθεια, αυτό είναι το τηλέφωνο το οποίο πρέπει να πάρει κανείς. Πρόεδρος. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε υποψήφιο επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ και όλους όσοι συμμετείχανε. Λήξη της ακρόασης.